Uh, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Περιμένω συναδέλφους, ελπίζω να έρθουν. Σήμερα είναι έτσι καλλιώς η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Συμβαίνουν αυτά. Χαίρομαι ιδιαίτερος που είμαι εδώ μαζί με τον Επίτροπο Αβραμόπουλο. Πρώτη φορά έρχεστε επισήμως στην ε, Επιτροπή μας. Είναι μεγάλη χαρά να σας συναντούμε για να μπορούμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων να σας ευχαριστήσω όμως για την παρουσία σας. Θα μας επιτρέψετε να δούμε κάποια σημεία στην ημερήσια διάταξη και να ε, μιλήσουμε μετά μαζί σας. Ε, θα συνεχίσω στα τελικά πρώτο σημείο, χαιρετώ τους ε, συναδέλφους και να θυμίσω ότι η κυρία Κάμερπερτ είχε ζητήσει να έχουμε μια σύντομη ενημέρωση στην αίθουσα για τον ε, τριμερή διάλογο για την ενιαία αγορά. Μπορούμε να το κάνουμε αύριο αυτό και κλεισμένο των θυρών ως τελευταίο σημείο, επειδή σήμερα έχουμε τόσα θέματα να δούμε στην εμείς διάταξη. Εάν συμφωνείτε. Μπορούμε λοιπόν με αυτή την ελαφρά αλλαγή να εγκρίνουμε την μέση διάταξη και να δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο. Πέτρα. Το ίδιο δεν είναι. Ωραία. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τα πρακτικά, θεωρώ είναι εγκεκριμένα στο δεύτερο σημείο και προχωρούμε. Μερικές ενημερώσεις. Πρώτα απ' όλα, διερμηνία σήμερα στις γλώσσες που βλέπετε. Γαλλικά, γερμανικά κλπ. Μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά. Η συνεδρία θα μεταδοθεί στο διαδίκτυο. Και να θυμίσω ότι έχουμε αύριο και την επίσκεψη και θα πάμε με λεωφορείο στον οργανισμό. Πριν δώσω τον λόγο στον Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, μου έχει ζητήσει τον λόγο ο συνάδελφος κύριος Γλέζος. Για δύο λεπτά. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ένα, ωραία. Και άλλη φορά μου έχει δοθεί η δυνατότητα να μιλήσω στην Επιτροπή μας ότι ο πολιτισμός είναι ταυτισμένος με τη δημοκρατία. Στην αρχαία Ελλάδα υπάρχει μια αλληλουχία λέξεων νοηματική και μορφολογική. Η μια πόλη όταν κατοικείται από πολίτες που ασκούν οι ίδιοι πολιτικοί το αποτέλεσμα είναι ο πολιτισμός. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε πολιτισμό εάν πολιτικοί δεν ασκούν οι ίδιοι οι πολίτες. Είναι ταυτισμένο το νόημα του πολιτισμού με τη δημοκρατία και τη σωστή της λειτουργία. Και το λέω αυτό για να πω ότι μου είναι αδιανόητο, όπως είπα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια και όπως θα τονίζω σε κάθε ευκαιρία ένας Ρωμαίος συγκλητικός στην ρωμαϊκή Σύγκλητο έλεγε «Χάνιμπαλ άντε πόρτας». Το ίδιο θέλω να πω και εγώ. Οι δανειστές έχουν φορέσει τη θηλιά να κρεμάσουν τον ελληνικό λαό χωρίς να σέβονται τη θέληση και τη βούληση του ελληνικού λαού ο ελληνικός λαός αποφάνθηκε. Δεν θέλω τα δάνεια, δεν θέλω τους δανειστές, θέλω να ελευθερωθώ. Αλλά οι δανειστές επιμένουν και γι' αυτό το λόγο δεν ε, ζητάω την γνώμη του ε, φίλου μου προσωπικού και συναδέλφου από παλιά στην πολιτική. Δεν ζητάω τη γνώμη του, όχι ούτε εκμεταλλεύομαι τη θέση του, θα το έλεγα οπωσδήποτε και αν ήταν ούτε θέλω να πάρει θέση θα κουβεντιάσουμε έπειτα το θέμα των, της μετανάστευσης. Αλλά θέλω να τονίσω ότι εάν μια επιτροπή σέβεται τον πολιτισμό Collega πρέπει Alexis, να σεβαστεί please. Because also you know that is out of the, this agenda, not the agenda of the European. Με συγχωρείτε, είναι εκτός της ημέρα για του Ευρωκοινοβουλίου, τη σημερινή συνεδρίαση. Σέβομαι, σέβομαι την ελεύθερη εκφρασή σα και την ελευθερία της ψυχής σας, αλλά Συμφωνώ και εγώ ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι αλληλέγγυα και υπάρχουν κανόνε δυστυχώ για τη σημερινή συνεδρίαση. Όλοι καταλάβαμε το νόημα του λόγου σα. Θα έλεγα να καλωσορίσουμε τώρα επισήμω τον Επίτροπο, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Όπω όλοι γνωρίζουν πολύ καλά, αρμόδιο για τη μετανάστευση, τι εσωτερικέ υποθέσει αλλά και του ε, πολίτε, στην τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαρά μας που σήμερα έχουμε αυτήν την συνάντηση, διότι κύριε Επίτροπε, για μας είναι πολύ σημαντικό και το θέμα του προπολογισμού ιδιαιτέρως, διότι τα δίκτυα των πολιτών από τα σχολεία και τους νέους μέχρι άλλες κοινωνικές, ε, άλλα κοινωνικά μορφώματα είναι πολύ σημαντικά στη συμμετοχή τους στον προπολογισμό. Αυτό επιτρέπει να ενισχυθούν οι αξίες οι κοινωνικές και της ηθαγένειας και που ισχύουν για τους Ευρωπαίους πολίτες και όσους διαμένουν στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικά λοιπόν αυτά για τον πολιτισμό. Θεωρούμε ότι το όλο θέμα είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό θέλουμε να ακούσουμε το τι θα μας πείτε, το πρόγραμμά σας Ξέρουμε ότι από την Γενική Διεύθυνση για την Παιδεία και την Πολιτισμό πέρασε στα δικά σας χέρια η αρμοδιότητα αυτή. Έχετε λοιπόν μια πολύ σφαιρικότερη ε, θεώρηση για τα θέματα αυτά και πολύ σημαντικά ζητήματα στο χαρτοφυλάκιό σας. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω το λόγο για τα θέματα αυτά, διότι στην περασμένη θητεία ζήσαμε κάπως δραματικά θα έλεγα την ε, περικοπή στο πρόγραμμα αυτό, 15%. 30 εκατομμύρια σχεδόν λιγότερο και γνωρίζουμε ότι στα διάφορα ελλείμματα του προγράμματος αυτού υπάρχει και μια γραμμή για την ε, αξιοποίηση και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Αυτό λοιπόν ξέρω ότι σας έχει απασχολήσει και το έχετε μελετήσει και θέλω να καταλάβω εάν η δέσμευση, οι διαδικασίες να γίνουν διαφανέστερες και αποτελεσματικότερες είναι κάτι που όντως μπορεί να πραγματοποιηθεί. Διότι υπάρχουν κάποια παράπονα από κάποιους συλλόγου, ενώσεις και ιδίως από τα σχολεία ότι η διδημοποίηση των σχολείων έχει, η αδερφοποίηση μάλλον των σχολείων έχει δυσκολευτεί. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα ευγνώμων για τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί Σα έχω συναντήσει στο Λουξεμβούργο, στη Ρώμη. Ξέρω πώ αγωνίζεστε για τα θέματα αυτά και προκειμένου να υπάρχει πραγματική αλληλεγγύη για ένα ζήτημα που καθόλου δεν απέχει από την ουσία του πολιτισμού. Διότι η ενσωμάτωση των μεταναστών ξεκινά πρώτα απ' όλα από το σχολείο, από τη διαδικασία τη εκπαίδευση. Ήδη τον Ιούλιο έχουμε προβλέψει συζήτηση για ένα θέμα και έκθεση της κυρία Γουόρτ για την πολιτιστική ποικιλομορφία και την εκπαίδευση και τα διαφορετικά πρότυπα και τις διάφορες προσεγγίσεις που μπορεί να υπάρχουν. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν οι διαδικασίε ενσωμάτωσης και εδώ νομίζω η συνεργασία μα μπορεί να είναι στενή. Υπολογίζουμε πολύ και σε εσά και στον Επιτροπό Ναύρατζιτ. Με αυτήν την εισαγωγή θα σας δώσω το λόγο για κανένα δεκάλεπτο και μετά μπορούν να παρέμβουν οι συνάδελφοι. Οι αξιολογότατοι συνάδελφοι που ξέρω ότι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Ε, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα μιλήσω τελικά, σήμερα αρκετά τόσο. Αγαπητοί βουλευτές, είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ σήμερα που τελικά μπορώ να μιλήσω στην δική σας Επιτροπή για την, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Να εκφράσω τις προσωπικές μου ευχαριστίες ε, στην Σίλβια Κώστα, την Πρόεδρο, για την ευγενική πρόσκλησή της όπως είπα πριν υπήρξε μια εισαγωγική συνομιλία μεταξύ μας όταν συναντηθήκαμε πρόσφατα στην Ρώμη. Το follow-up της συνάντησής μας στην Ρώμη θα είναι πολύ ε, διαφορετικό. Θα είναι μια συνάντηση στο Λουξεμβούργο, πολύ διαφορετική από αυτή που έχουμε εδώ. Ε, τι να κάνουμε. Και οι δύο θέλαμε λοιπόν αυτή η συνάντηση να γίνει νωρίτερα. Αλλά όπως γνωρίζετε ήταν πολύ δύσκολο, αν όχι δεν ακούγεται η γερμανική μετάφραση. Ακούτε τη γερμανική μετάφραση παρακαλώ, όχι. Όπως είπα πριν, και οι δύο θέλαμε αυτή η συνάντηση να γίνει νωρίτερα. Όμως ήταν αδύνατο και πραγματικά ζητώ την κατανόησή σας γι' αυτό, γιατί πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο το πρόγραμμα. Όλοι γνωρίζετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας. Τους τελευταίους μήνες υπήρχε επίγουσα ανάγκη να ανταποκριθούμε σε αυτά τα φοβερά γεγονότα που έχουν ταράξει την Ευρώπη. Έχουμε την κρίση με τη μετανάστευση στην Μεσόγειο και όλα αυτά τα ζητήματα που ζητούσαν την άμεση και πλήρη προσοχή της Επιτροπής. Όλα αυτά τα γεγονότα που μόλις ανέφερα είχαν ε, άμεση επίπτωση στους Ευρωπαίους πολίτες και ξεκάθαρη επίπτωση, διότι οι πολίτες πραγματικά νοιάζονται για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και θέλουν να απολαμβάνουν αυτά τα δικαιώματα μέσα σε μια ασφαλή κοινωνία οι πολίτες δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι οι άνθρωποι που ζητούν προστασία θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και πεθαίνουν στη Μεσόγειο. Το να αντιμετωπιστούν λοιπόν αυτές οι προκλήσεις και να, να υπάρξει ανταπόκριση στις ανησυχίες ε, των ε, Ευρωπαίων πολιτών παρουσιάσαμε την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια και την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την ε, μετανάστευση. Αυτή ήταν η απάντηση της Κομισιόν. Ε, ε, έχοντας εξηγήσει αυτά, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αυτό το θέμα των Ευρωπαίων πολιτών είναι ένα από τα πιο σημαντικά και λόγω των πρόσφατων εξελίξεων πραγματικά γίνεται μία από τις προτεραιότητές μας. Πρέπει να επανέλθουμε στις αρχές ε, ε, αυτού του ονείρου που δημιούργησε την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή όλα φαίνεται ότι τίθενται υπό αμφισβήτηση τα δικαιώματα και η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια ε, στην ουσία αποτελούν την ουσία της ανάγκης και της επιτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. όλο και μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων επικρίνουν σήμερα το ευρωπαϊκό εγχείρημα και τις βασικές, τα βασικά του επιτεύγματα, για παράδειγμα το Σέγγεν και το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών και των αγαθών, το οποίο πραγματικά εγώ ε, θεωρώ ότι ως μέρος της ε, ε, γενιάς των οραματιστών ε, που είδαν ε, ανθρώπους να περιμένουν ουρές στα σύνορα ε, απαντώ ότι όχι, δεν θα επιτρέψουμε. Δεν επιστρέψουμε σε αυτές τις μέρες. Αυτές που οι νέοι μας δεν έχουν βιώσει. Σήμερα η ξενοφοβία, ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός οδηγούν όχι μόνο σε απαράδεκτες συμπεριφορές, αλλά και σε εγκληματικές και τρομοκρατικές επιθέσεις. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα? πώς να αλλάξουμε τις αντιλήψεις και πώς να δημιουργήσουμε ένα θετικό αφήγημα. Ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της δουλειάς είναι το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες» που είναι στη δική μου ευθύνη. Οι στόχοι του προγράμματος αυτού είναι πραγματικά επίκαιροι και όχι μόνο μέσα στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, αλλά και σε πολλές ε, πολιτικές ε, που έχει στην αρμοδιότητά της η Κομισιόν. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν σήμερα που έχω την ευκαιρία να το συζητήσουμε μαζί και να σας παρουσιάσω τις πρώτες μου σκέψεις, αλλά κυρίως να ακούσω τις δικές σας. Παρόλο που ο προπολογισμό είναι σχετικά μετριοπαθής για αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτε είναι ουσιώδε σε επίπεδο περιεχομένου. Υποστηρίζει δραστηριότητε που καλύπτουν την συμμετοχή των πολιτών στα κοινά σε όλη την Ευρώπη, κάτι που θα έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Προσφέρει χρηματοδότηση για τα ευρωπαϊκά έργα, τα project και τις ε, πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε μία εμβάθυνση της κοινή κατανόησης, της ιστορικής μνήμης και του διαπολιτισμικού διαλόγου, της αλληλεγγύης, τη συμμετοχή των πολιτών της κοινωνίας μάλλον και ε, σε τοπικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα από πέρυσι. Στη Γαλλία υπήρξε το έργο που ονομαζόταν ε, επιτυχία, success και ε, αποτελεί το από ένα δίκτυο νέων από διαφορετικά πολιτισμικά, κοινωνικά υπόβαθρα και οικονομικά υπόβαθρα που ζούσαν σε πολυπολιτισμικές και μειονεκτικές γειτονιές και ζητούσαν από τους Ευρωπαίους πολίτες να συνεισφέρουν στην ανατροπή των ε, ρατσιστικών, λαϊκιστικών και ξενοφοβικών τάσεων στην Ευρώπη και να προωθήσουν τις ουσιώδεις αξίες, τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια υπήρξαν σκέψεις σχετικά με τη ε, συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στα κοινά, στην πολιτική ζωή, στην τοπική κοινωνία. Ε, υπήρχαν σκέψεις ε, για την πολυπολιτισμικότητα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ούτω καθεξής. Είχαμε και συναντήσεις μεταξύ Ευρωπαίων και εθνικών πολιτικών Μιλήσαμε για το κάψιμο των βιβλίων από τους Ναζί και για την απαγόρευση κάποιων λογοτεχνικών έργων κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Στάλι. Ε, αυτό ε, έγινε μια, έγινε μια συζήτηση γι' αυτό για τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την ε, Ρωμανία και τη Σλοβενία. Η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, των πολιτών, των ενδιαφερόμενων και των όσων λαμβάνουν τις αποφάσεις στην ευαισθητοποίηση και στη συζήτηση για τις αξίες της Ευρώπης είναι κομμάτι της ελευθερίας έκφρασης στην Ευρώπη. Για να δούμε τώρα την ευρύτερη εικόνα. Το 2014 το πρόγραμμα Ευρώπη για τους ε, πολίτες συγχρηματοδότησε 412 project από 31 χώρες ε, και σε, αυτό το, σε αυτά τα προγράμματα συμπεριλήφθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες. Έγιναν αδελφοποίησεις πόλεων, δίκτυα πόλεων, project της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και για τη μνήμη της Ευρώπης. Όπως επίσης δόθηκαν και επιχορηγήσεις σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δρούν τους θεματικούς τομείς ε, στους οποίους ε, στοχεύει το πρόγραμμα. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτά τα project ε, τα εφαρμόζουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφοσιώσει τη ζωή τους ολόκληρη στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Έτσι λοιπόν οι πολίτες αναπτύσσουν ενεργό, ενεργά την ευρωπαϊκή ιδέα και προωθούν την αξία της συμμετοχής και της κοινή δράσης για τη δημιουργία, την οικοδόμηση μιας καλύτερης Ευρώπης. Αυτό το πρόγραμμα πριν καν έρθει στη δική μου αρμοδιότητα ως ε, Επιτρόπου Μετανάστευσης έπρεπε να αντιμετωπίσει την, τον κοινωνικό διάλογο και τις ανησυχίες των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών, γιατί στην ουσία η διαχείρισή του γίνεται από κάτω προς τα πάνω, με την προσέγγιση bottom-up. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα και την ευκαιρία, θα έλεγα, να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να κάνουν κάποια project που σχετίζονται με τη μετανάστευση, την οικονομική κρίση και τις κοινωνικές επιπτώσεις τους. Είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι η ανάγκη να δοθεί νέα, νέος ρυθμός σε αυτό το πρόγραμμα είναι κάτι που ε, απαιτείται ξεκάθαρα. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Έχουμε ε, τακτικές ε, ε επικοινωνίες με τα think tank και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και από αυτή την άποψη θα έπρεπε να αναφέρω ότι αυτή ακριβώς τη στιγμή, παράλληλα με τη δική μας συνεδρίαση, οι υπηρεσίε της Κομισιόν και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες ε, κάνουν στην ουσία την πρώτη τους ε, συνάντηση για τον κοινωνικό διάλογο της φετινής χρονιάς. Θα ανταλλάξουν λοιπόν απόψεις για το ποιες θα είναι οι προτεραιότητες του 2016. Ομοίως με ενδιαφέρει να ακούσω και τις δικές σας προτάσεις και ιδέες, οι οποίες θα είναι πραγματικά πολύτιμες για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε το πρόγραμμα εργασίας για το 2016. Θα το υποβάλουμε στη Συμβουλευτική Επιτροπή, στην Επιτροπή Διαβούλευσης ε, το Σεπτέμβρη για να μπορέσουμε να το εγκρίνουμε πριν τα τέλη του έτους. Αγαπητοί φίλοι, όταν μιλάμε για την ε, η ηθαγένεια, αναφερόμαστε στην ευρωπαϊκή ηθαγένεια και στα δικαιώματα που παίρνει ο κάθε πολίτης μέσα από τις συνθήκες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ηθαγένεια λοιπόν έχει πολλά πολύτιμα δικαιώματα, το δικαίωμα κίνησης και ελεύθερης εγκατάστασης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα δικαιώματα πολιτικής συμμετοχής στις ευρωπαϊκές και δημοτικές εκλογές και προστασία κατά των διακρίσεων. Η ευαισθητοποίηση λοιπόν και η ενίσχυση ως προς αυτό το θέμα είναι ένας από τους βασικούς ρόλους της Κομισιόν. Του χρόνου η Επιτροπή μας θα παρουσιάσει την τρίτη έκθεσή της για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Η έκθεση αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται υπό την ηγεσία του Επιτρόπου Τζούροβα συγγνώμη, και η, πρόεδρος, η, η πρόοδος που έχει δημιουργηθεί ε, πραγματικά θα αντανακλάται στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες, ε, λοιπόν, ε, στην ουσία ξεκινά να ψάχνει και για συμπληρωματική σχέση με άλλες πολιτικές αυτό έχω ζητήσει από τις υπηρεσίες μου ως πρώτο βήμα. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, αγαπητή Επιτροπή, αυτή η η ηθαγένεια είναι ένα κοινό αίσθημα το, που έχουμε όλοι ότι ανήκουμε σε μια Ευρώπη με κοινέ αξίες. Ήτανε πραγματικά η λογική, η λογική που οδήγησε στην πρόοδο την Ευρώπη είναι μια αρχή που παραμένει και δίνει νόημα στην όλο και στενότερη ένωση. Είναι λοιπόν χαρά μου και τιμή μου που είμαι υπεύθυνο για αυτό το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες και που έχω τακτικό διάλογο με την Επιτροπή σας. Για άλλη μια φορά λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και φυσικά δίμονο να υπάρξει μια επικοδομητική συζήτηση και μια ε, σημαντική συνεργασία στο μέλλον σε αυτόν τον πολύ σημαντικό ε, χώρο, την ε, κοινή μας πατρίδα, την Ευρώπη. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Εκτιμούμε ιδιαίτερος την αναφορά σας στην στενή διασύνδεση των προγραμμάτων για την Εθαγένεια και τη σχετική πολιτική με τα θέματα που αποσχολούν την Επιτροπή Πολιτισμού. Το πολιτιστικό διάλογο, την εκπαίδευση και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την τοποθέτηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στον πυρήνα όλων αυτών των ε, ζητημάτων πρωταγωνιστούν και κάποιες φορές και με ερνητικό ρόλο εκπροσωπούν τις διαφωνίες και τις συγκρούσεις της κοινωνίας τις δυσκολίες ενσωμάτωσης αλλά κάποιες φορές και με τη θετική συνεισφορά του προγράμματος που αναφέρατε. Ένα πρόγραμμα που για σας είναι πολύ σημαντικό και με, τον απαραίτητο, με την απαραίτητη πρικοδότηση και τις προτάσεις του συναδέλφου Ντρογεύσκη που ελπίζουμε να επηρεάσουν θετικά ε, καθ' ο εισηγητής, ελπίζουμε να συμβάλλουμε και εμείς αυτή την προτεραιότητα. Είναι, μια, ε, είναι συμβολικής αξίας το να επενδύσουμε στο πρόγραμμα αυτό. Και τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. η κυρία Κάμερπερ, Τρούπελ και άλλοι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που σήμερα είσαστε εδώ για να συζητήσετε μαζί μας στην Επιτροπή Πολιτισμού για ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα την Ευρώπη των Πολιτών. Εδώ στην Επιτροπή μας νομίζω ε, πραγματικά ε, δεν έχουμε καταλάβει γιατί στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα μειώθηκαν ε, η χρηματοδότηση για αυτό το πρόγραμμα όπως και από τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε γιατί πραγματικά αυτό το πρόγραμμα είναι ένα από τα λίγα με τα οποία μπορούμε άμεσα να έχουμε επαφή με τους πολίτες και να υπάρχει κατανόηση για τις βασικές αξίες της Ευρώπης, να τις προωθήσουμε και να τις ενισχύσουμε. Λοιπόν, Καλό ε, όταν έχουμε κρίσεις και τέτοια πράγματα αρνητικά που διαβάζουμε παντού, ε, δεν είναι καλό και είναι αντιπαραγωγικό τα θετικά να τα ε, κουρεύουμε έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει πραγματικά να υπάρχει η απέτηση να γίνει από την πλευρά της Κομισιόν ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να υπάρχει μια καλή κατανομή πορών σε αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, μια ερώτηση για την Κομισιόν. Υπάρχει έλλειψη σε επίπεδο διοικητικό και ε, υπάρχουν πάρα πολλά ε, ε, έγγραφα που πρέπει κανείς να συμπληρώσει για αυτό το πρόγραμμα αυτό. Το ακούμε από τις οργανώσεις, από εταιρικές αποτερίες. Γενικά λένε ότι υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία για τις αιτήσει και υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις για να μπορεί κανείς ε, να λάβει έγκριση για ένα έργο μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, μάλιστα για αυτούς που είναι εθελοντές. Ε, υπάρχουν ε, λοιπόν απαιτήσει για να έχουν κάποιους συμβούλους, όμως δεν μπορούν. Είναι σχεδόν αδύνατο. Ζητούν λοιπόν να δουν τι θα γίνει γιατί ας πούμε και η ανταλλαγή μεταξύ δύο-τριών ε, μικρότερων εταίρων είναι πολύ δύσκολη και δεν μπορούν αυτές οι οργανώσεις σήμερα να αντέξουν πολλά οικονομικά. Πρέπει λοιπόν να δούνε αν ε, κάποιο κομμάτι αυτού του προϋπολογισμού θα μπορούσε να δοθεί για τις μικρότερες εταιρικές σχέσεις. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που ε, σήμερα βρίσκεστε εδώ για να συζητήσετε μαζί μου. Πραγματικά συντάσσομαι πλήρως με αυτά που είπε και η προλαλή σας. Ε, πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε καθόλου και πραγματικά θα έπρεπε να αμυνθούμε στεναρά έναντι του γεγονότος ότι αυτό το πρόγραμμα δεν έχει πλέον τόσα κονδύλια. 200 ε, ε, εκατομμύρια ευρώ για έξι χρόνια σε 28 κράτη-μέλη πραγματικά είναι μια σταγόνα στον ωκεανό για ένα τόσο σημαντικό ε, και απαιτητικό πρόγραμμα με όλα όσα πρέπει να αντιμετωπίσει. Συντάσσουμε λοιπόν με την ερώτηση αυτή. Ακούμε συνεχώς ότι όλοι και, οι μεγάλοι παίρνουν χρηματοδότηση και αυτό είναι λάθος προσέγγιση. Νομίζω ότι σε αυτό το τομέα που ε, έχει να κάνει με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στα κοινά. Μιλάμε ε, για την Ευρώπη των ανθρώπων. Πρέπει οι, άνθρωποι μέσα στην Ευρώπη να έρθουν πιο κοντά ο ένας στον άλλον και πραγματικά αυτό μόνο με τα μικρά έργα μπορεί να γίνει, όχι τόσο με τα μεγάλα. Ε, είναι σημαντικά και τα μεγάλα, αυτό δεν το συζητάμε, όμως είναι ο καιρός και οι μικρές οργανώσεις ε, που πραγματικά έχουν μεγάλη ε, αφοσίωση και συμμετοχή ε, να μην αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις δυσκολίες ε, να ε, πληρούν τις προδιαγραφές για τα έργα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κάποιες σκέψεις στην Κομισιόν για τις κατευθυντήρες γραμμές του προγράμματος κυρίως από την εμπειρία που έχετε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να συλλέξετε, αν μπορούμε να τις αναθεωρήσουμε κάπως ώστε να διευκολυνθεί, να γίνει πιο απλό ε, σε επίπεδο διαδικασιών το πρόγραμμα. Να μην ε, ε, έχουμε μόνο τους μεγάλους όπως σας είπα, αλλά να έχουμε και μικρότερα έργα που θα χρηματοδοτούνται τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο να ε, βλέπουμε αυτή τη συνεργασία που έχει τόσες μεγάλες επιπτώσεις να ευωδώνεται. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Ε, υπάρχει δυνατότητα ενδεχομένως ε, και για άλλα προγράμματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έργα που συγκεκριμένα μπορούν να χρηματοδοτηθούν τα οποία στην ουσία προωθούν αυτή την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας να τα ενισχύσουμε. Αυτά δηλαδή που ε, έχουν παρόμοιο στόχο, άλλα προγράμματα, άλλα project. Και ίσως ε, τα χρήματα που λείπουν από τη μία πλευρά να τα αντισταθμίσουμε με την άλλη αυτό. Υπάρχει τουλάχιστον συνοχή στις ερωτήσεις. Η κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο για την ομιλία του. Συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες» είναι σημαντικό. Από την άλλη πλευρά, πολλές είναι οι επικρίσεις που έχουν, επικρίσεις που έχουν ασκηθεί. Μειώθηκε ο προϋπολογισμός, αλλά αυτό ίσως είναι ένα ανόητο εγχείρημα από τη στιγμή που θέλουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να επικοινωνούν, να ξεκινούν με νέα project, με νέα σχέδια. Ερωτώ λοιπόν, είστε έτοιμοι να βρείτε επιπρόσθετες δυνατότητες μέσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο για το πρόγραμμα αυτό. Και επίσης, στην επόμενη, στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο <clears throat> θα ασκήσετε μεγαλύτερη πίεση αυτό το πρόγραμμα να έχει περισσότερη ορατότητα και περισσότερο προϋπολογισμό. Γιατί ξέρετε πολλοί υπέβαλαν αίτηση για το πρόγραμμα αυτό και απορρίφθηκαν. Μας μιλήσατε για τις επιτυχίες, αλλά ξέρουμε ότι όλο και περισσότερα έργα απορρίπτονται. Και αυτό δεν είναι καθόλου διαφήμιση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά δεν ενδιαφέρεται. Και αυτό είναι κάτι αρνητικό για εμάς και για την ε, κοινή ευρωπαϊκή ιδέα. Από εκεί και πέρα και ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν, λαμβάνουν υπόψη, δεν λαμβάνονται υπόψη έργα που έχουν να κάνουν με την Αφρική. Θέλουμε να υπάρξει ένα σύστημα μπόνους για το κόστος που μπορεί να υπάρχει ε, για την μεταφορά, για τις μετακινήσεις, έτσι ώστε να έχουν οι χώρες τη δυνατότητα να συνεργαστούν. Είναι ένα θέμα που αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ Βορρά και Νότου και Ανατολής και Δύσης. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ίσως καλύτερα να απαντήσετε σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις πρώτα και μετά στους επόμενους τρεις. Παρακαλώ, Επίτροπε. Ήξερα ότι τέτοιες ερωτήσεις έπρεπε να περιμένω. Επιτρέψτε μου όμως ευθύς ε, εξ αρχής να πω το εξής. Και στις τρεις ερωτήσεις ο βασικός πυρήνας ήταν τα χρήματα, ο προϋπολογισμός και δεν είστε οι μόνοι που παραπονιέστε για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το εξής ό,τι έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό είναι και στα δικά σας χέρια. Γιατί είστε συνομοθέτες εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως, ας συμφωνήσουμε σε κάτι. Ας κάνουμε μια συμμαχία σήμερα. Θα σας παρουσιάσω κάποιες προτάσεις και θα τις στηρίξετε. Εφικτό παράδειγμα του πώς μπορούμε να δουλέψουμε μαζί. Και είπα ότι είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε όλα αυτά τα προγράμματα, όλα αυτά τα έργα. Ξέρετε, ορισμένοι στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι αυτό που κάνουμε εδώ, που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, είναι πράγματι πολύ σημαντικό. Και ε, είναι όμως σημαντικό, αλλά δίνουν προτεραιότητα ενδεχομένως σε άλλα ζητήματα. Και καταλαβαίνετε ότι για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός και να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες της Ευρώπης σήμερα και για να συνδεθούμε με αυτούς οι οποίοι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποφάσισαν να δημιουργήσουν την Ευρώπη, προκειμένου λοιπόν να επιστρέψουμε στις ρίζες μας, η πρόκληση υψώνεται μπροστά μας. Πρέπει να καλλιεργήσουμε την ευρωπαϊκή συνείδηση και πρέπει να ξεκινήσουμε να χτίζουμε την Ευρώπη από τη βάση της κοινωνικής πυραμίδας, από κάτω προς τα πάνω. Επομένως, ναι, χρήματα χρειάζονται, συμφωνώ με αυτό και θα το στηρίξω αυτό, γιατί όλα αυτά είναι πολύ κοντά στη δική μας πολιτική φιλοσοφία για το μέλλον της Ευρώπης. Τώρα, για το διοικητικό βάρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει φτιάξει τα σημεία επαφής ε, της Ευρώπης για τους πολίτες. Έτσι ώστε σε αυτά τα κέντρα να διαδίδεται η πρακτική πληροφόρηση για τις δραστηριότητες, για τις δυνατότητες χρηματοδότησης, για όλα. Ως προς το νεπίγοντα χαρακτήρα της εφαρμογής του προγράμματος «Η Ευρώπη για τους πολίτες», η ACA, έχει θεσπίσει ένα σύγχρονο σύστημα management διοίκησης για να γίνεται σωστή διαχείριση του προγράμματος επιτόπου, ε, απρόσκοπτη και εύρυθμη. Βλέπετε λοιπόν ότι πλησιάζουμε τις απόψεις σας. Ίσως και τα μικρά προγράμματα είναι πολύ σημαντικά για μας όχι μόνο τα εμβληματικά προγράμματα, τα ευρύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο συνάδελφος ή συνάδελφος Κάρσον. Όμως βγαίνει. Έχατε το λόγο. Μάουρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω απολύτως με την αντίληψη του αγαπητού Επιτρόπου, τον οποίο και καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Και θα ήθελα να αξιοποιήσω το γεγονός ότι ανακοίνωσε το ενδεχόμενο συμμαχίας μεταξύ της Επιτροπής μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να πω ότι από πλευράς μου θα σας παράσχω κάθε δυνατή στήριξη σε κάθε πρωτοβουλία που θα παρουσιάσετε κύριε Επίτροπε. Βεβαίως θα τις εξετάσω όλες τις προτάσεις τις συγκεκριμένες πολύ προσεκτικά, εάν και εφόσον τις παρουσιάσετε. Σε κάθε περίπτωση. Ε, θα ακολουθήσω τη γραμμή σκέψης που υιοθέτησαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Γιατί είχα την ευκαιρία να γνωρίσω το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες» γιατί ήμουν εισηγητής για τον προϋπολογισμό για το 2013 και τότε είχα, πα, είχα συζητήσει με διαφόρους εμπλεκόμενους φορείς ε, για την εκπόνηση της έκθεσής μου τότε και πρέπει να σας πω ότι είχα σημειώσει ότι ορισμένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποβάλλουν, δεν παρουσιάζουν κανένα πρόγραμμα, κανένα έργο για το Europe for Citizens, για την Ευρώπη, για τους πολίτες, για το πρόγραμμα αυτό. Πολύ περίεργο μου φαίνεται αυτό και παράδεκτο σχεδόν. Δηλαδή σε καιρούς κρίσης όπου πλήττεται η ευρωπαϊκή συνείδηση και η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το να υπάρχουν κράτη-μέλη που να μην υποβάλλουν προς έγκριση ούτε ένα σχέδιο ούτε ένα έργο στο πρόγραμμα αυτό ε, λοιπόν επαναλαμβάνω ότι μου φαίνεται εξαιρετικά περίεργο. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς άλλη εξήγηση γι' αυτό. Ωστόσο, οι χαμηλές προσδοκίες για την επιτυχία υπάρχουν. Αυτή είναι η αιτία που κάνει κάποιον να μην υποβάλει αίτηση, να λειτουργεί αποτρεπτικά όλη αυτή η διαδικασία. Σκέφτεται κανείς ότι και να υποβάλει την αίτηση, να υποβάλει πρόταση για το πρόγραμμα ε, δεν θα ε, εγκριθεί. Και αυτό λειτουργεί ε, απογοητευτικά και αποτρεπτικά. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλη εξήγηση για την κατάσταση αυτή. Και όντας ο προϋπολογισμός τόσο χαμηλός, πρέπει να στηρίξουμε οποιοδήποτε μέτρο θα βελτίωνε την κατάσταση. Επομένως, επαναλαμβάνω, στηρίζω την άποψη και την πρόταση του Επιτρόπου και θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τις συγκεκριμένες, επαναλαμβάνω, συγκεκριμένες προτάσεις που έχει να υποβάλει γιατί σίγουρα πολλές από αυτές μπορούμε να τις στηρίξουμε όλοι. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Μάουρα. Ο συνάδελφος Γλέζος. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην Πρόεδρο για το γεγονός ότι προσκάλεσε εδώ για συζήτηση τον αρμόδιο επίτροπο για τα κέρια αυτά θέματα. Όντως, το ερώτημα η Ευρώπη των πολιτών. Δηλαδή στην ουσία σοβαρολογούμε ή παίζουμε με τις λέξεις. Η Ευρώπη ανήκει στους πολίτες της ή η Ευρώπη ανήκει στο ΝΑΤΟ και στο εμπορικό ΝΑΤΟ που ετοιμάζεται τώρα με σκοπό να παρασέρνεται από τις Ηνωμένε Πολιτείες και να μην είναι αυτοδιοικούμενη, αυτόνομη και αυτοδιοίκητη. Τι θέλω να πω με αυτό. Στην αρχαία Ελλάδα η λέξη Ευρώπη είναι κάτι το καταπληκτικό. Είναι το αντιμέτωπο του κύκλοπα. Ο κύκλοπς τι ήταν. Σύνθετη λέξη από τις λέξεις κύκλος και το ουσιαστικό του ρήματος ορά ορό όψ οπός. Δηλαδή ο κύκλοπας είχε ένα μάτι γιατί δεν μπορούσε να δει τα πράγματα πολυδιάστατα. Έπρεπε να τα δει μονοδιάστατα. Μέσα σε ένα κύκλο έβλεπε τα πράγματα, από όπου και ξεκινήσει το ίδιο σημείο θα φτάσει. Η Ευρώπη όμως, το αντίθετο, είναι η πολυδιάστατη αντίληψη, ο ανοιχτομάτης, ευρύς και πάλι όψ όπως, του ρήματος ραωρό, που σημαίνει ότι βλέπω τα θέματα πολυδιάστατα. Ρωτάω, η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει τα θέματα πολυδιάστατα ή μονοκόμματα τα βλέπει και καταπιέζει τους πολίτες. Εδώ είναι βασικό το θέμα. Όσους και συναντάω και όσους και αν βλέπω και όσους και αν μιλάω μου λένε δεν θέλω να αποφασίζει άλλος για μένα. Λέω αυτό είναι το πρόβλημά σου μονάχα. Λέει είναι. Υπάρχει λέει κι άλλο, λέω βεβαίω. Όχι μονάχα δεν θέλω να αποφασίζει άλλος για μένα αλλά θέλω να αποφασίζω και εγώ συμμετέχοντας στα κέντρα λήψη των αποφάσεων. Αυτό γίνεται στην Ευρώπη. Λυπούμε που θα το πω, δεν είναι κρυφό πράγμα, ο φίλος μου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος το γνωρίζει πολύ καλά, ξέρει ότι δεν του χαρίζομαι και σε τίποτα, υπηρετεί σήμερα τις απόψεις του Γιούγκερ, ο οποίος θέλει την Ευρώπη κάτω από τις δικές του διαταγές. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Υπηρετώντας τα αμερικανικά κεφάλαια της ολιγαρχίας υπηρετώντας το κεφάλαιο. Λοιπόν, να μην κοροϊδευόμαστε, η Ευρώπη πρέπει να γίνει η Ευρώπη των πολιτών, συμμετέχοντας οι πολίτες στα κέντρα λήψη των αποφάσεων. Όσο για το άλλο θέμα της μετανάστευσης, θα αναφέρω ότι στην αρχαία Ελλάδα πάλι υπήρχε ένα προσωνύμιο στον Δία, ο ξένιος Δίας. Δηλαδή, ο Ξένιος Δίας ήταν η πλευρά του Δία που προστάτευε τους ξένους. Όσους προσέφευγαν προς άσυλο σε οποιοδήποτε μέρος και ιδιαίτερα στους ναούς. Σήμερα το κύμα των μεταναστών έρχεται και μας ζητάει καταφύγιο και εμείς το αρνούμαστε. Και μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν νεκροί από τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφύγουν στην Ευρώπη. Θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη και ζητάνε άσυλο στην Ευρώπη. Και τα βόρεια κράτη αντιμετωπίζουν τους μετανάστες της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας τα αντιμετωπίζουν. Λύστε εσείς το πρόβλημα μόνοι σας. Πώς να το λύσουμε μόνοι μας. Πώς να το λύσουμε μόνοι μας. Εμείς βέβαια πιστοί στην αρχή του ξένου Ουδία, πιστοί στην αρχή του ασύλου θα προστατεύσουμε τους μετανάστες ό,τι και αν λέει η υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά δεν είναι Ευρώπη αυτή όταν αντιμετωπίζει έτσι το θέμα. Έχω κουβεντιάσει επανειλημμένα με τον Επίτροπο. Κολέγα Γκλέτος, can you... στο τέλος με πιάσετε. Λοιπόν, έχω κουβεντιάσει επανειλημμένα, στο έχω πει και η βασική αιτία είναι τα αίτια. Αν δεν προκαλούσαμε συγκρούσεις εμείς για τα πετρέλαια στις χώρες εκείνες δεν θα υπήρχαν μετανάστες. Εάν εμείς δεν συνεχίζαμε την υποταγή των χωρών που είχαμε προηγούμενα ως απικίες, δεν θα υπήρχαν μετανάστες. Λοιπόν, να δούμε τη βασική αιτία και να λύσουμε τα ουσιαστικά ζητήματα και λυπούμε τον Δημήτρη που θα υπερασπιστεί το Γιούγκερ πάλι και όλη τη μαφία, το λέω έτσι καθαρά, των ολιγαρχών γύρω από αυτό το θέμα, ενώ ξέρω ότι έχει άλλες απόψεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Γλέζο. Η ε, συνάδελφος Σοντρόβα. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, να σας ευχαριστήσω για την ε, ομιλία σας και να σας βεβαιώσω ότι είμαι πρόθυμη να στηρίξω τον προϋπολογισμό Ευρώπη για τους πολίτες. Έχω μεγάλη εμπειρία με συναλλαγές με τους πολίτες, με διάφορες κοινότητες, με τους φοιτητές. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Νέων. Ένα πρόγραμμα εξαιρετικά ενδιαφέρον, ένα παράδειγμα που δείχνει πώς μπορεί να λειτουργήσει το κοινοβούλιο και πώς μπορούν να προετοιμαστούν τα προγράμματα από τους νέους, από τους φοιτητές, για τους φοιτητές. Φοιτητές που δεσμεύονται, που θέλουν να χτίσουν μια κοινή Ευρώπη και συνάδελφε Γλέζο πρέπει να πω ότι δεν αμφιβάλλω. Το μέλλον της Ευρώπης είναι για τις νέες γενιές, για αυτές πρέπει να το φτιάξουμε. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό η Ευρώπη για τους πολίτες πρέπει να είναι πολύ πιο ανοιχτό, ευρύ και να συμπεριλαμβάνει τις νέες γενιές, τους φοιτητές. Είμαι λοιπόν πρόθυμη να στηρίξω την ενίσχυση αυτού του προγράμματος, ώστε να στηριχθούν τα προγράμματα για τους νέους, τους φοιτητές που θέλουν να προσφέρουν, να συμμετάσχουν ε, στην ε, ζωή, στο βίο της Ευρώπης. Αυτό είναι το μέλλον μας και αυτό οφείλουμε να πράξουμε. Δυστυχώς, ε, είναι βέβαιοι ότι το πρόγραμμα αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους Νέους, δεν λαμβάνει στήριξη από το πρόγραμμα που αναφέραμε. Αντιθέτως θα έλεγα, δεν ισχύει αυτό και ελπίζω να αλλάξει σύντομα αυτό που συμβαίνει. Σας ευχαριστώ για την αφοσίωση στο σκοπό σας. Ευχαριστούμε ο λόγος στην κυρία Ward. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι. με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω πόσο ανοιχτό αντιμετωπίζεται τα θέματα αυτά επίτροπε με μια επιτροπή πολύ ανανεωμένη και πολύ σφρυγιλή πρέπει να πω. Είμαστε μια ιδιαίτερα δραστήρια επιτροπή πολιτισμού. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στα παιδιά. Είμαι μέρος, μέλος ε, ομάδας προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών και εδώ στο Κοινοβούλιο και εκτός. Ε, ε, πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στη σημασία των πολιτών των ίδιων, ιδίως των πολιτών του μέλλοντος, η άμεση συμμετοχή ή δυνατόν στο έργο μας εδώ στο Κοινοβούλιο ε, θα είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει, διότι το δικό τους το μέλλον να διαμορφώνουμε. Ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να ξέρω εάν η συμμαχία που θέλετε να έχουμε μαζί, εσείς και εμεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει τα παιδιά και του νέου. Και να προτείνω μια πολύ άμεση κίνηση που θα μπορούσατε να κάνετε το καλοκαίρι φέτο. Μαζί με κάποιου ε, από την κοινοβουλευτική μου ομάδα συμμετέχω σε μια έκτακτη εβδομάδα δραστηριοτήτων για παιδιά και νέου από όλη την Ιφίλιο, στην Ελβετία, την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου συγκεκριμένα. Δεν θα έλεγα να έρθετε ω εκεί, αναγκαστικά, αλλά αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα ή να είχαμε συνομιλία μέσω Skype, ώστε τα παιδιά και οι νέοι να έχουν άμεσα συζήτηση μαζί σας. Νομίζω θα τους έκανε πάρα πολύ καλό να σας ε, απευθύνουν το λόγο και να σας ε, μιλήσουν για τα θέματα που τους αποσχολούν. Και δύο συγκεκριμένε ερωτήσεις. Έχουμε σοβαρές ανησυχίες για τα δικαιώματα των παιδιών, ιδίως των ε, παιδιών μεταναστών. Πρώτα απ' το άρθρο 3 της χάρτα των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των παιδιών λέει ότι όλες οι ενέργειες προς παιδιά από ε, δημόσιους φορείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή δικαστήρια ή διοικητικούς φορείς ή νομοθετικούς φορείς θα πρέπει να σκοπεύουν στην ύψιστη προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά των μεταναστών, ασχέτως από το καθεστώς που έχουν οι γονείς τους ως προς την ιδιότητα του μετανάστη. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύονται τα δικαιώματα όλων των παιδιών μεταναστών με όλες τις μορφές πολιτικής και δράσης που μπορεί με την ε, διεκπαιρέωσή τους να έχουν κάποια επίδραση στα παιδιά. Επίσης η κράτηση των παιδιών δείχνει ότι έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ψυχική και σωματική τους υγεία, ακόμη και αν πρόκειται για πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα. Η Επιτροπή λοιπόν του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των παιδιών και το Συμβουλίο της Ευρώπης έχουν καταστήσει σαφές ότι παρά ασχέτως μάλλον με το καθεστώς ε, του παιδιού ή του γονέα ε, είτε το παιδί έχει έρθει συνόδευτο είτε με τους γονείς του δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται κράτηση παιδιού. Πώς μπορείτε να ενθαρρύνετε τα κρατη μέλη να εφαρμόσουν ε, αυτό το νόμο όπως την οδηγία των περιεπιστροφών και σε συμφωνία με αυτά τα διεθνή πρότυπα για τα δικαιώματα των παιδιών. Ευχαριστούμε για αυτή τη του παρατήρηση, Τζούλη. Να δώσω το λόγο και στην κυρία Τρούπελ, διότι έχει μια συγκεκριμένη ερώτηση και μετά θα σας δώσουμε το λόγο, Επίτροπε. Ευχαριστώ. Ένα ερώτημα δεν απαντήσατε κύριε Επίτροπε. Το θέμα του συστήματος μπόνους για υψηλό κόστος μεταφοράς και ταξιδίου μετάβασης. Το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες» πολύ συχνά ασχολείται με προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται σε ένα μικρό κύκλο, δύο-τρεις περιφέρειες γειτονικές. Αν θέλουμε να είναι πραγματικά ευρωπαϊκό θα πρέπει να εμπλέξει πολύ πιο απομακρυσμένες περιφέρειες και άρα τα έξοδα μετάβασης θα πρέπει να ε, ε, επιδοτούνται με κάποιο βαθμό, να στηρίζονται. Έχετε κάτι να πείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ενδιαφέρον θα ήταν, δεν θέλω να σας πιέσω να απαντήσετε τώρα, θα έχουμε και άλλε ευκαιρίες, ποια θα είναι η ισορροπία τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των τοπικών φορέων και των σχολείων. Διότι έχω την εντύπωση ότι η διάσταση των σχολείων κάπως ε, αποδυναμώνεται. Ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει, κάποιοι φορεί, ε, αλλά τι θα γίνει με τα σχολεία. Και αύριο έχουμε μια συνάντηση με τον οργανισμό ΕΝΣΑ για από που είναι από την αιγίδα του Επιτρόπου Ναύρατσιτ, εκεί μπορεί να λάβουμε κάποιες απαντήσεις. Θα μπορούμε να εμβαθύνουμε δηλαδή εκεί για την υλοποίηση του όλου κανονισμού. Ευχαριστώ. Let me start by the last... Καταρχάς να ξεκινήσω με το τελευταίο ερώτημα. Δεν απάντησα πριν γιατί ε, ρωτούσα να ενημερωθώ περί τίνος πρόκειται. είναι λίγο τεχνικό να το επαληθεύσω και να επανέλθω με συγκεκριμένη απάντηση. Τώρα, ως προς το εξής σχόλιο, ότι κάποια κράτη-μέλη δεν υποβάλλουν έργα για να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό να σας υπενθυμίσω ότι η η ποιότητα ενός έργου είναι και πρέπει να παραμείνει το βασικό κριτήριο για την επιλογή του. Από το 2007 μέχρι και το 2008, πέντε χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία και Πολωνία, ήταν αυτές οι οποίες κατά 80% υπέβαλαν αιτήσει για έργα που θα ενταχθούν ή θα εντάσσονταν στο πρόγραμμα. Το 2013 το ποσοστό είχε πέσει στο 54% αυτών των πέντε χωρών. Τώρα, όταν έπεσε το μερίδιο της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας, το, το αντίστοιχο της Ιταλίας και της Ουγγρανίας αυξήθηκαν σημαντικά. Η Ιταλία και η Ουγγαρία ε, υπέβαλαν πάρα πολλές αιτήσει και τις περισσότερες τις υπέβαλαν το 2013 και το 2014. Τώρα, ορισμένα νέα κράτη μέλη γνώρισαν σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Σλοβακία, Ρουμανία και Σλοβενία είναι αυτές που κυρίως υπέβαλαν αιτήματα για ένταξη στο πρόγραμμα. Τώρα η Εστονία, η Λετωνία και η Λιθουανία τριπλασίασαν τον αριθμό των αιτήσεων καθ' όλη τη διάρκεια αυτή της περίοδου. Ωστόσο, οι αιτήσει από την Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν σε αριθμό. Άρα θα μπορούσε κανείς να διαβάσει μια τάση ε, των πιο πεπειραμένων, να το πω έτσι, κρατών μελών να απομακρύνονται από μικρά έργα και να πλησιάζουν ε, περισσότερο μεγάλα έργα ε, βάθους και μακράς χρονικής διάρκειας. Τα εθνικά σημεία επαφής θα πρέπει να μας βοηθήσουν να μας βοηθήσουν να προβάλλουμε, να προωθήσουμε και να κάνουμε την επικοινωνία του προγράμματος αυτού, η Ευρώπη για τους πολίτες. Και ελπίζω όλα τα κρατημέλη να μας δώσουν ένα σημείο επαφής. Και άλλωστε το Εθνικό Σημείο Επαφής θα βοηθήσει τα έργα μικρού μεγέθους να ανταποκριθούν καλύτερα στα προαπαιτούμενα, στις απαιτήσει του προγράμματος «Η Ευρώπη για τους πολίτες». Και θα πω δύο λόγια στα ελληνικά για να απαντήσω ε, στον Μανώλη Γλέζο. Οπότε σας παρακαλώ να βάλτε τα ακουστικά σας. Αγαπητέ μου Μανώλη, αν και δεν ανήκουμε στην ίδια γενιά, ξέρεις ότι σε τιμούμε πολύ στην Ελλάδα. Για μας είσαι ένα σύμβολο και πάντοτε σε ακούμε με πάρα πολύ προσοχή αλλά θα με επιτρέψετε να σα πω ότι σε ορισμένα πράγματα δεν συμφωνώ. Εγώ ανήκω στη γενιά εκείνη που έβγαινε στου δρόμου και αγωνιζόταν ω φοιτητή για μια Federal Europe, για μια ομοσπονδιακή Ευρώπη. Mm. Πριν από λίγο ανέφερα κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών και είναι μια προσωπική εμπειρία. Όταν φοιτητής θα να κάνουμε Interrail, οι παλιότεροι το ξέρουν αυτό, με 150 δολάρια μπορούσε να ταξιδεύει με τρένο από τη μια γωνιά τη Ευρώπη στην άλλη. Και διψάγαμε τότε να γνωριστούμε μεταξύ μα οι νέοι τη Ευρώπη. Στο πρώτο μου ταξίδι σε ηλικία 19 χρονών, με backpack και μένοντα σε hostels τη εποχή εκείνη, και έχοντα γνωρίσει κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα πάρα πολλού Ευρωπαίου, διεπίστωσα ότι ήταν το όνειρο μια ολόκληρη γενιά. Όταν όμω γύρισα στην Ελλάδα πήγα και άλλαξα διαβατήριο. Γιατί το διαβατήριό μου είχε τόσες πολλές φραγίδες που δεν χώραγε πλέον καμία. Σήμερα μπορώ να ταξιδεύω ακόμα και με το δίπλωμα οδηγήσεως. Γι' αυτό σας είπα πρωτήτερα ότι πρέπει να προστατεύσουμε αυτή τη μεγάλη κατάκτηση. Και όσο περισσότερο γνωρίζονται οι λαοί και οι πολίτες μεταξύ τους, τόσο περισσότερο βρίσκει έδαφος η προσπάθεια που κάνει αυτή η Επιτροπή και που είναι στην βάση της συλλογική μας προσπάθειας να ξαναφέρουμε την υπόθεση της ευρωπαϊκής συνείδησης στο προσκήνιο. Και εκεί που θα συμφωνήσω μαζί σου είναι ότι άλλαξαν οι προτεραιότητες. Αλλά η Ευρώπη σταδιακά και αργά μεν προχωράει. Μόνο που ο στόχος πρέπει να παραμείνει, από την δική η πολιτική της ενοποίηση για να ενισχύσει περισσότερο την αυτονομία της και να μπορεί να διαδραματίσει τον παγκόσμιο ρόλο που της αναλογεί. Αλλά ποτέ να μην απομακρυνθεί από τους πολίτες. Δεν θα συμφωνήσω επίσης μαζί σου τώρα που τον γνωρίζω καλύτερα για τον πρόεδρο Γιούγκερ, οποίο συμπτωματικό είναι και πολύ καλό φίλο τη Ελλάδο και νομίζω το ετοιμάει και το εκτιμάει ο ελληνικό λαό. Και τον τελευταίο καιρό κάνει μεγάλε προσπάθειε για να βρει τον περίφημο αυτό δίκαιο συμβιβασμό ώστε να λυθεί το πρόβλημα και να προχωρήσει μπροστά. Είναι ίσω από του τελευταίου μεγάλου Ευρωπαίους σαν και εκείνους που γνώρισε η δική σου γενιά μετά τον πόλεμο και η οποία ακριβώς είχε το όνειρο να φτιάξει μια Ευρώπη χωρίς σύνορα, ειρηνική, δημιουργική, προοδευτική. Τότε ήταν που ελέγχθη ποτέ πόλεμος πια. Και απευθύνομαι σε σένα γιατί εσύ τον βίωσε τον πόλεμο. Και γι' αυτό σου είπα ότι είσαι σύμβολο όχι μόνο της Ελλάδα, αλλά και άλλων λαών γιατί όλοι ξέρουν το μεγάλο σου επίτευγμα της εποχής εκείνης αλλά μην αδικούμε ούτε τις τότε γενιές, ούτε όμως και τις σημερινές. Και θα έλεγα και κάτι άλλο, μιας και το ανέφερες. Προέκταση της Ευρώπης είναι η Αμερική. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Τον ευρωπαϊκό πολιτισμό υιοθέτησε, από Ευρωπαίους μετανάστες φτιάχτηκε και σήμερα εκατομμύρια Ελλήνων, Ιταλών αποτελούν την δύναμη αυτής της κοινωνίας. Το αντίθετο πρέπει να γίνει να καλλιεργηθεί ακόμη περισσότερο ο διάλογο και να εγκατασταθεί περισσότερη εμπιστοσύνη για όλα τα θέματα που από κοινού πλέον αντιμετωπίζουμε, πολλά εκ των οποίων έχουν να κάνουν με το χαρτοφυλάκιό μου. Και αναφέρομαι και σε θέματα ασφάλεια και σε θέματα μετανάστευση. Το όνειρο πρέπει να είναι το ίδιο. Έκανα σκόπο να τα πω αυτά και πήρα και εγώ λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί τον άλλο τον βλέπω τον εκτιμώ, τον αγαπώ, αλλά καμιά φορά ξυπνάει μέσα ο επαναστάτης των 18 του χρόνων όταν τότε κατέβαζε την αριστική σημαία από την Αγρόπολη. Αλλά αυτή η εποχή πέρασε, σήμερα και με τους Γερμανούς συμβιώνουμε μαζί και ένας λαός που πρόκοψε πολύ, κατάφερε πολλά μέσα από τα συντρίμια και την ταπείνωση σήμερα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και θέλουμε και εμείς από όπου και αν βρισκόμαστε να είμαστε όλοι στην κοινή, στο κοινό μέτωπο και μια καλύτερη, πιο συνεκτική, πιο ενωμένη Ευρώπη που να μας οδηγεί το κοινό όραμα το οποίο ξεκινάει, το επαναλαμβάνω, από την συνείδηση των πολιτών. Και γι' αυτό είπα ότι αυτή η Επιτροπή χρειάζεται στήριξη και θα την έχει, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, μια και ένα μεγάλο κομμάτι της έχει να κάνει με το χαρτοφυλάκιό μου, διότι πάει κοντά στο σημείο από όπου ξεκινάει ή αν θέλετε όπου χρειάζεται να ξαναγεννηθεί το όραμα της νέας μεγάλης μας πατρίδας της Ευρώπης. before about migrants' children. Μίλησα για τα παιδιά των μεταναστών, αλλά ας μιλήσουμε γενικότερα για τα παιδιά, είτε είναι δικά μας της Ευρώπης, είτε τα παιδιά των μεταναστών. Όλα παιδιά είναι. Οπότε θα συμφωνήσω πολύ με τις πρωτοβουλίες σας και ναι, δέχομαι την πρόσκλησή σας. Θα είμαι εκεί είτε αυτοπροσώπος, είτε χάρη στις νέες τεχνολογίες μέσω του Skype αλλά με έναν και μόνο σκοπό, να σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε αμύωτες τις προσπαθίες σας, που είναι τρομερά σημαντικές, για να γίνει πιο ανθρώπινος ο κόσμος μας. Η προστασία των παιδιών είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων μου. Κατά την ακρόαση με τους συναδέλφους σας της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ πριν 9 μήνες, ανέλαβα δέσμευση να εργαστώ για αυτό το σκοπό. Και ήδη έχουμε αρχίσει να έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα. Εάν δείτε την, το νέο θεματολόγιο για τη μετανάστευση, θα δείτε ότι αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στα παιδιά των μεταναστών. Ας ελπίσουμε τα κράτη-μέλη να μας βοηθήσουν. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολλά ακούγονται σε θεωρητικό επίπεδο τι τελευταίε ημέρε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Πριν από λίγα λεπτά άκουσα επικριτικά σχόλια για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ρώτησε ο Μανώλης Γλέζος τι κάνει η Ευρώπη. Ε, και εγώ αντεπιτίθεμαι και λέω τι κάνουν τα κρατημέλη. Εγώ έχω υπάρξει υπουργό ε, επανειλημμένο στο παρελθόν και όποτε ερχόμουν στι Βρυξέλλε και να προσπίσω τα εθνικά μου συμφέροντα. Δεν σκεφτόμουν ούτε εδρούσα ω Ευρωπαίο. Τώρα είμαι από την άλλη πλευρά, στην άλλη όχθη του ποταμού, αλλά ο ποταμό αυτό βρίσκεται στην ίδια χώρα. Ξέρω λοιπόν πώ αισθάνονται τα κράτη-μέλη, ε, πώ ε, σκέφτονται και δρούν, αλλά ξέρω και πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί μπορούν να δράσουν. Αν λέμε διαρκώ λοιπόν για την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σίγουρα έχουν διαφορετική προσέγγιση, αλλά πρέπει να του δείξουμε εμεί τον δρόμο. Να δούμε πώ μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να ε, ενεργούμε κατά τον ίδιο τρόπο. Επίση, γιατί κρατούσα σημειώσει. Επίσης να τονίσω ότι και τα δύο προγράμματα που ανέφερα στις αρχικές μου παρατηρήσεις συμπεριλαμβάνουν τα παιδιά. Όμως, ως γενική παρατήρηση, να πω κάτι παραπάνω. Η συμμετοχή των νέων γενικώ είναι κάτι που έβρισκε σύμφωνο. Όχι μόνο φοιτητέ, όλοι, ε, ενώσεις, σύλλογοι, τα πάντα. Τις τελευταίους εννέα μήνες, ίσως είναι δική μας ευθύνη, αυτό που είδα είναι ότι, ίσως να πρέπει να βρούμε είδα ότι η νεολαία δυστυχώς κρατιέται μακριά μας. Ίσως ε, εξαιτία των όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, λόγω χάρη ανεργία. Δεν μας εμπιστεύονται. Δεν μας εμπιστεύονται όπως οι προηγούμενες γενιές. Αλλά πρέπει να πάμε εμείς προς το μέρος τους. Και να τους θυμίσουμε ότι το πρόγραμμα αυτό η Ευρώπη για τους πολίτες είναι πολύ σημαντικό. Πολύ ακριβές και πολύ διαφανές. I don't have else to, to, say for the moment. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο προς στιγμή, εκτός αν κάτι ξέχασα, αλλά είμαι στη διάθεσή σας. Ό,τι θέλετε μπορώ να απαντήσω. Ευχαριστώ. <laughs> Uh, uh, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία σας και για τις απαντήσεις σας. Υποσχεθήκατε προηγουμένως ότι οι τεχνικές λεπτομέρειες μπορεί και να απαντηθούν ε, γραπτός, αλλά και αύριο η συνάντησή μας είναι πολύ σημαντική και θα έχουμε τις απαραίτητες ε, πληροφορίες. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Επιτροπό Αβραμόπουλο για την ε, επίσκεψή του. και οι συνάδελφοι σίγουρα σημειώνουν όσα είπε με προσοχή. Όλοι μοιραζόμαστε τη ίδιο όνειρο για την Ευρώπη και εγώ στην ίδια περίπου γενιά ονειρεύτηκα μια διαφορετική Ευρώπη και θέλουμε να μην μετατραπεί σε φιάλτη η Ευρώπη θα πρέπει να είναι μια εναλλακτική και ενώπιον των διώξεων, των θρησκευτικών πολέμων, των μετακινήσεων πληθυσμών, δεν θα πρέπει να δείξουμε εχθρική στάση. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν θα πρέπει να ενισχυθεί όχι μόνο λόγω της συμβολικής του αξίας, αλλά επειδή και στην πράξη λειτουργεί. Ε, το παίρνουμε λοιπόν πολύ σοβαρά το πρόγραμμα αυτό και εσείς επίσης πάρτε σοβαρά τις προτάσεις μας για προτεραιότητες, ε, το πρόγραμμα αυτό για την Ευρώπη των Πολιτών και βεβαίως τη συνάδελφος Δρογεύσκα που ασχολείται με τον προπολογισμό. Το θέμα αυτό ήδη το έχουμε επισημάνει και ελπίζουμε στις διαπραγματεύσεις σας με το Συμβούλιο να βρείτε κοινέ προτεραιότητες. Πιστεύω ότι από αυτή την άποψη μπορούν να υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες και να συνεργαστούμε, διότι αμφιβολία δεν υπάρχει ότι η Ευρώπη για τους πολίτες σημαίνει για τα δικαιώματα της ηθαγένειας, αλλά της ε, κοινωνικής διάστασης, της ε, εκπαιδευτικής, των ε, κοινών αξιών και της ε, συνύπαρξης. Νομίζω λοιπόν θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες και θα είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε στην Επιτροπή Πολιτισμού, Παιδείας και Νέων. Σας ευχαριστώ ξανά. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους. Ξέρω ότι έχετε ενημένες υποχρεώσεις. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πολύ, Επιτροπέ. Colleghi, Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, συνάδελφοι, σημείο 5 της σημερινής διαταξής, Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό Έτο 2016. Το συζητούσαμε και προηγουμένω. Ε, να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον προπολογισμό ήδη ε, στις 27 Μαΐου υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ σύντομα γνωρίζετε ότι για το 2016 η Επιτροπή Πολιτισμού πρέπει να εγκρίνει τρεις θέσεις, τρία βήματα δηλαδή, ε, γνωμοδοτήσεις για τον προπολογισμό που μετά ε, αποστέλλονται στην Επιτροπή Προπολογισμού που διαπραγματεύεται εκ μέρους του Ευρωκοινοβουλίου. Σήμερα το απόγευμα έχουμε εδώ τον κύριο Φερνάντες που είναι ο εισηγητής εκ μέρους του Ευρωκοινοβουλίου για τον προπολογισμό του 2016 και είναι μια καλή ευκαιρία για να έχουμε μια σοβαρή συζήτηση για το θέμα αυτό. Ε, η συνάδελφος Ντρογεύσκα έχει αναλάβει το θέμα αυτό εκ μέρους της Επιτροπή μα. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα λοιπόν γι' αυτό. Και αύριο θα έχουμε ψηφοφορία για την πρώτη από τις τρεις ε, γνωμοποιήσεις αυτές στην Επιτροπή μας και με το αποτέλεσμα θα δώσουμε εντολή στην, στον ε, εισηγητή για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών θεσμών. Στην Ολομέλεια η έκθεση αυτή θα περάσει από, ε, το, στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Το δεύτερο βήμα είναι όταν στην συνεδρία της Επιτροπής τον Ιούλιο θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες για τον ίδιο τον προπολογισμό τις ε, παρατηρήσεις δηλαδή και τους αριθμούς. Σήμερα ψηφίζουμε ε, για το σχέδιο προπολογισμού που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Μαΐου. Υπάρχουν και τα θέματα που μας αφορούν εδώ πέρα βεβαίως, ε, πολιτισμός, παιδεία και επικοινωνία. Η προθεσμία για την των απολογιών είναι 30 Ιουνίου. Κανονικώς οριζόντια εντολή θα αποδοθεί στον εισηγητή τον Ιούλιο για να μπορέσει εφόσον γίνουν γνωστές οι αντιπροτάσεις του Συμβουλίου να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις και με το Συμβούλιο βάσει και των όσων θα μας πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τον Σεπτέμβριο το τρίτο βήμα, το τρίτο step με τη δική μας συμβολή για την τελική μορφή της έκθεσης για τον προπολογισμό το 2016. Αυτή θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου ε, και έτσι θα ολοκληρωθούν οι διάλογοι μεταξύ των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Είναι ο πρώτο προπολογισμό που υποβάλλει η Επιτροπή Juncker και θα πρέπει να συγχαρούμε τους συνοδέλφου που συμμετείχαν και στήριξαν τη συμμετοχή της Επιτροπής ε, Πολιτισμού και Παιδείας όχι μόνο γιατί συμπεριέλαβαν τα θέματά μας μεταξύ των προτεραιοτήτων, αλλά και τις ε, νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά θέματα που μας απασχολούν και θα συνεχίσουν να τα παρακολουθούν. Σε αυτή τη φάση θα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Στρογεύσκα και σε όσους άλλους θελήσουν να συμμετάσχουν. Παρακαλώ. Tak, E, Κυρία Πρόεδρε, να σα ευχαριστήσω και πάλι, διότι έχετε κάνει τη δουλειά μου εδώ πιο εύκολη. Επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι εδώ στην ουσία έχουμε να κάνουμε με τρία έγγραφα. Το πρώτο θα συζητηθεί σήμερα και θα ψηφιστεί αύριο. Υπάρχει μια σειρά τροπολογιών και υπάρχει και ένα πρόβλημα με τις ε, προθεσμίες. Και αυτό το τρίτο έγγραφο, το ψήφισμα, θα ισχύει για το 2006. Να σας θυμίσω ότι όσον αφορά στις ε, προθεσμίες, όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, έχουμε χρόνο μέχρι την 30η Ιουνίου. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 14 Ιουλίου. Αυτό υπόθηκε ήδη, όμως η νομοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού αυτή τη στιγμή ακόμη είναι υπό επεξεργασία και δεν υπάρχει ε, καταληκτική ημερομηνία. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους πάντες για τη συνεργασία σε, αυτό το σχέδιο γνωμοδότητης υπάρχουν ε, γύρω στις 30 τροπολογίες. Προσπαθήσαμε και επιτύχαμε να ε, υπάρξει συμβιβασμός και οι υπεύθυνοι των τροπολογιών με χαρά συζήτησαν και ε, ήρθαν ο ένας πιο κοντά στον άλλον ως προς τις θέσεις τους. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Στρόπελ και άλλους για τις τροπολογίες, ε, τους κύριους ε, Μάρα κυρία Ζωηντρόβα, για την πολύ καλή εικόνα πραγματικά. Έχουμε ε, συμφωνήσει για κάποιες βασικές προτεραιότητες εδώ. Καταρχάς για την πρόθεση και υποστήριξη του προγράμματος Erasmus Plus, Erasmus Sin. Υπάρχει μια γενική συμφωνία επί αυτού. Επίσης, είμαστε υπέρ της προώθησης του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Υπάρχει και γενική συμφωνία και σε επίπεδο αντίδρασης προς αυτό, αλλά και σε επίπεδο συστάσεων. Και το τρίτο πρόγραμμα είναι η Ευρώπη για τους πολίτες που ήδη συζητήθηκε. Η χρηματοδότηση έχει ελαφρώς αυξηθεί για το 2016 σε σχέση με το τρέχον έτος. Υπάρχει προφανώς κάποιος λόγος να χαρούμε. Οπότε ε, βλέπετε ότι υπάρχει μια προφανής πρόοδος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια δεν έχει εμπριστατώσει τα ποσά που στην ουσία είναι διαθέσιμα και την κατανομή αναπρόγραμμα. Θα έχω τις πληροφορίες ε, και μόλις τις έχω θα σας τις ε, παραθέσω. Τώρα για τις τροπολογίες σχετικά με το προϋπολογισμό του 2016 υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες. Πρώτον, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ειδικότερα το Erasmus ΣΥΝ, Δημιουργική Ευρώπη, πρέπει να έχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση, τα απαραίτητα κονδύλια, όμως αυτά τα κονδύλια πρέπει να κατανέμονται χρονικά με το σωστό τρόπο, έτσι ώστε οι δαπάνες να συνάδουν με τις προβλέψεις. Αυτό που έχει βελτιωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πολιτική επικοινωνία και η προώθηση αυτών των δραστηριοτήτων στι τρίτες χώρε, αλλά και στα κράτη-μέλη όπου ε, εκτελούνται αυτά τα πολιτιστικά έργα, τα project. Όπως το Euroland Sin. Υπάρχει η γενικότερη συμφωνία επίσης για την ανάγκη να υποστηρίξουμε τους νέους ανθρώπους, ειδικότερα τους νέους δημιουργούς και καλλιτέχνες, αυτούς που εργάζονται στον τομέα του πολιτισμού σε μια σειρά ε, προγραμμάτων και έργων για τον πολιτισμό. Είμαστε υπέρ επίσης της υποστήριξης των μικρότερων project υπό το πρίσμα του, από την γενικότερη έννοια του πολιτισμού, γιατί προωθούν την ποικιλομορφία στην Ευρώπη. Υπήρξε λοιπόν μια ενδιάμεση ε, επισκόπηση όλων αυτών των μικρότερων project και φαίνεται ότι υπήρξε μείωση στον πολιτισμό και σε αυτά τα μικρά project γενικότερα. Για να δούμε τώρα τις ε, προθεσμίες. Υπάρχει από την Κομισιόν ένα πρόγραμμα και θέλουμε να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε γιατί ε, για να καταφέρουμε να βγάλουμε αυτά τα χρονικά περιθώρια θα πρέπει να δουλεύουμε και Σάββατα και Κυριακές. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 14 Ιουλίου όπως σας είπα και αυτό θα είναι πριν την πιλωτική αξιολόγηση και την προπαρασκευαστική εργασία από την πλευρά της Κομισιόν. Αυτό προφανώς είναι προβληματικό, αλλά έχει και κάποια θετικά στοιχεία, διότι ίσως η δική μας ψηφοφορία τελικά να επηρεάσει αυτά που θα συμβούν στην Κομισιόν. Ε, πολλές φορές λοιπόν υπάρχει φως στην άκρη του τούλνελ, δεν είναι όλα μαύρα. Υπάρχουν λοιπόν τρία, τρεις κατηγορίες, τρεις ομάδες. Αυτή που ασχολείται με την ψηφιοποίηση και την προώθηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας κινηματογράφων, δεύτερον εκπαίδευση και κινητικότητα των νέων, ειδικότερα ε, στις ε, περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στα σύνορα και τρίτον η προώθηση ε, της, ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Έπρεπε από κάθε πολιτική ομάδα λοιπόν να γίνει μια πρόταση για να μπορέσουμε να αποφύγουμε κάποιες ομάδες να έχουν αποκλειστικά ε, κάποια θέματα. Να τονίσω ότι όλα αυτά τα project σχετίζονται ξεκάθαρα με μικρότερα που με τη σειρά τους προωθούν κάποιες πλατφόρμες ας πούμε για τα φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ευρώπη. Δεν είναι ακριβά και βελτιώνουν την επικοινωνία από τη δική μας πλευρά. Αυτά κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τη συνεργασία, ειδικότερα για τις συμβαστικές τροπολογίες που πραγματικά θα ικανοποιήσουν πλήρως όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Ευχαριστούμε συνάδελφε Στρογεύσκη για τη δουλειά σας και την υπόσχεση να παρακολουθήσετε με προσοχή όλα αυτά τα θέματα. Μου φαίνεται όμως πολύ σωστό να ε, προσέξουμε και πώς θα αντιδράσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Η προτεραιότητά σας πάντως είναι προτεραιότητες που συμμεριζόμαστε. Να δώσω πρώτα απ' όλα το λόγο στον συνάδελφο Μόργανο που είναι σκιώδης εισηγητής. Αυτή τη στιγμή έχουν το λόγο οι σκιώδης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με όσα μάλλον μας είπε ο εισηγητής και τον ευχαριστώ για την ακριβέστατη ε, παρουσίαση του θέματος. Προφανώς γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς τι μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε εξαιτία των σοβαρών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης από την οποία φαίνεται με δυσκολία βεβαίως να βρίσκουμε κάποια διέξοδο, αλλά οι θετικές ακόμα ε, συνέπειες, τα θετικά αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν αισθητά και από τους Ευρωπαίους πολίτες. Δίνω έμφαση σε αυτό, διότι γνωστή η στατικική έμφαση της ανάκαμψης ε, και της ε, Ανάπτυξης σε συνδυασμό με την απασχόληση και την Επιτροπή μας. Αυτό είναι ένας σκοπός και ένας στόχος του εισηγητή αλλά και όλων μας. Δηλαδή να προστατεύσουμε τις ε, δεσμεύσεις πτώσεων για την άσκηση του προπολογισμού του 2015, για το Erasmus ΣΥΝ, για την Ευρώπη της Δημιουργίας και την Ευρώπη των Πολιτών. Όπως γνωρίζουμε στο σχέδιο προπολογισμού όπως υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το θυμήσαν αυτό οι συνάδελφοι, η Επιτροπή ε, Κουλτ είναι υπεύθυνη για τις ε, για 85 γραμμές του προπολογισμού, μεταξύ των οποίων στα, ε, στους τίτλους 15, εκπαίδευση και πολιτισμός και 16 επικοινωνίας. το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορούν τα τρία πολυετή προγράμματα ε, ως προς την πρικοδότησή τους, τα οποία μόλις ανέφερα. Αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη προβολή και είναι τα πλέον δημοφιλή μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Τα οποία λοιπόν έχουν μεγάλη πολιτική σημασία στη διαδικασία λήψη αποφάσεων που τώρα ξεκινά και θα μα οδηγήσει στην έγκριση του προπολογισμού για το 2016. Αυτά τα λέω διότι εδώ υπάρχουν παρεμβάσεις που προβλέπουν επιμέρους επιδοτήσεις οι οποίες θα πάνε κατευθείαν σε πρόσωπα και οργανισμούς με άμεση δηλαδή σχέση και συμμετοχή της Ένωσης από την Ένωση στα χέρια των ε, αρμοδίων. Κατά τον ίδιο τρόπο και όπως ε, με σαφήνεια το εξέφρασε στην ε, γνωμοδότησή του ο συνάδελφος, εισηγητής, για τον τριμερή διάλογο και την εντολή του θα πρέπει να επαγρυπνούμε για το θέμα των απλήρωτων λογαριασμών. Το είπαμε αυτό, είναι ένα θέμα άκρος ευαίσθητο, διότι και το λέω αυτό και επιμένω, οι προβλέψεις για πληρωμές ε, στα επόμενα σχέδια προπολογισμού θα πρέπει και αυτό το λέω ε, με επιμονή, ε, θα πρέπει να γίνουν μακροπρόθεσμα και με διάρκεια, όχι μόνο για τον προπολογισμό του 2016, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις πληρωμές που δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρουμε ότι πρέπει να δούμε αν υπάρχει πραγματική κάλυψη, πλήρης ή μερική και αν οι αριθμοί που μετά παρουσιάζονται ε, βάσει των όσων θέλουμε για το 2016 εάν θα βασιστούν στα όσα έγιναν το 2015 εάν θα βασιστούν σε απλήρωτους ε, λογαριασμούς σε ποσά που δεν καταβλήθηκαν αυτό έχει σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για τους πολίτες αλλά και τις οικογένειες που όλα αυτά αφορούν Βλέποντα λοιπόν τα στοιχεία του υπολογισμού, επιτρέψτε μου δύο στοιχεία στα οποία ήθελα να εμείνω, διότι τα ε, μελέτησα και τα βρήκα βάσει των διαθέσιμων στοιχείων. Υπάρχει αύξηση του λειτουργικού κόστους που ξεπερνά το 5% και νομίζω ότι είναι σημαντική η αύξηση 120 εκατομμυρίων για το Erasmus Plus αλλά υπάρχει και αύξηση στις πληρωμές 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το θέμα είναι λοιπόν να καταλάβουμε ποια θα είναι ε, αυτά που ε, θα ε, δοθούν ως προτεραιότητα. Τα ακούσαμε και από τον Επίτροπο αυτά στα θέματα για τα οποία είναι αρμόδιο, αλλά πρέπει να δούμε τι θα κάνει και η Γενική του Διεύθυνση. Η Δημιουργική Ευρώπη επίση, η Ευρώπη τη Δημιουργία. 15 εκατομμύρια ε, αύξηση με πληρωμές 50 εκατομμύρια και για την Ευρώπη των πολιτών αύξηση 1 εκατομμύριο με αύξηση των πληρωμών 7 εκατομμύρια. Το είπα και προηγουμένως. Θεωρώ ότι ο αριθμός που ε, περιλαμβάνει ο προπολογισμός ως προς τα προγράμματα αυτά δείχνει και το τι ε, προβολή θέλουμε να δώσουμε το πολιτικό προσκήνιο στις πραγματικές μας ενέργειες και στα προγράμματα που παρουσιάζουμε. Ως προς τους αριθμούς αυτούς λοιπόν δεν μπορώ να μην πω προσωπικώς ότι με απασχολεί το γενικότερο πλαίσιο. Ξέρουμε ότι κοιτάζοντα το μέλλον, θα πρέπει να σκεφτούμε τι γίνεται και με τα πιλωτικά προγράμματα. 25 εξ αυτών και το πρόβλημα είναι να καταλάβουμε πώς θα απαντήσουμε ε, τι λύσεις θα βρούμε για τα 25 αυτά προγράμματα ανάλογα με την ποιότητα και ούτω καθεξής αλλά και επειδή εδώ ε, κάποιο κριτήριο πρέπει να υπάρχει. Είναι επίσης σημαντικές οι 8 προπαρασκευαστικές δράσεις και επειδή ακόμα βρισκόμαστε στην πρώτη φάση της διαδικασίας στο Κοινοβούλιο, υπάρχει η συνήθεια στην Επιτροπή Κούλτ να καταλήγουμε σε μία θέση ομοφωνίας, την οποία όλοι να τη συμμερίζονται. Όχι απλώ ότι δηλαδή εγκρίνουμε τουλάχιστον για τα προγράμματα και τι δράσει τη δική μα αρμοδιότητα, διότι είναι σημαντικά όχι μόνο για μα αλλά και για του πολίτε μα. Αυτό σήμερα είναι ένα στοιχείο που πρέπει να υπογραμμιστεί και από πολιτική άποψη να στηριχθεί. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε για αυτήν την ανάλυση. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε προτεραιότητε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, για τι πληρωμές. Πληρωμέ που σέρνουμε εδώ και τρία χρόνια και ε, μία ενημέρωση ε, που να είναι τουλάχιστον συνεπής. Η συνάδελφος Τρούπελ. Ήθελα απλώς να αναφέρω κάποια σημεία. Το πρώτο είναι ότι θυμάμαι, πιστεύω ότι οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες θα πρέπει να παραμείνουν στρατηγικής σημασίας εντός του ε, ΕΦΣΥ, οπότε θα πρέπει να το επιδιώξουμε εμείς ως Επιτροπή θέλουμε να έχουν στατηγικό ρόλο η, επι... παιδεία και ο πολιτισμός εντός του ΕΦΣΥ. Και θα πρέπει όλες οι επιτροπές να επιδιώξουν μεγάλες επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό και για αυτόν τον προπολογισμό είναι το θέμα του, Oiron, του Euronet, ότι εδώ χρειάζεται μια συμφωνία ε, που έχει από όλους ε, εγκριθεί να υπάρχει περισσότερη ε, χρηματοδότηση εδώ για το Erasmus Plus για το Erasmus ΣΥΝ θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει εδώ με τον προπολογισμό, με την αύξηση που ήδη υπάρχει. Θέλουμε να χρηματοδοτηθούν τα μικρά προγράμματα, ιδίω και μέσω των περιφερειακών ταμείων. Υπήρχε ανέκαθεν τάση στην Επιτροπή να, πηγαίνει για να δίνει προτεραιότητα στα μεγάλα προγράμματα, διότι για διοικητικού λόγου αυτό είναι ευκολότερο. Όμω από τη δική μα την Σκόπια θα πρέπει να κοιτάξουμε να καλύπτουμε στο δυνατόν περισσότερους ανθρώπου, Οπότε έμφαση έχει δοθεί στο ότι θέλουμε να ε, ε, χρηματοδοτηθούν μικρά προγράμματα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ε, και τα δικτυωμένα προγράμματα τα έχουν σημαντικές συνέπειες. Να θυμίσω ότι το Ευρώπη για τους πολίτες έχει μεγάλη σημασία γιατί ακριβώ υπάρχουν πολλά λησυνδεόμενα προγράμματα. Αυτό είναι πάντοτε μια σημαντική λεπτομέρεια. Άλλοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο ή να κλείσουμε εδώ τη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάτι να μας πει, υπάρχει κάποιος που θέλει να παρέμβει ή είναι ακόμα στη φάση των πρώτων διαβουλεύσεων και... Η Επιτροπή μας θα παρακολουθήσει με ιδιαίτερη προσοχή ε, τα όσα συμβαίνουν και θα προασπιστεί τον προπολογισμό για τον πολιτισμό, την παιδεία και τους νέους. Θα αφογκραστούμε όλες τις εξελίξεις. Θα είναι χρήσιμο αυτό και για τον εισηγητή μας. Θέλετε το λόγο, ε, κύριε Στρογεύσκη. <laughs> Ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί, αγαπητά μέλη της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Σημειώσαμε τα διάφορα σχόλια σε σχέση με τις δημοσιονομικές προοπτικές. Βλέπετε ότι αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για το Erasmus Sin και το 20 Europe. Αυξήθηκαν οι πιστώσεις οι διαθέσιμες για την πληρωμή και αυτό οφείλεται στο ότι μπορέσαμε να ε, μειώσουμε τις καθυστερούμενες ληξιπρόθεσμες, καθυστερούμενες οφειλές. Και ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να χρηματοδοτήσουμε τα νέα έργα του 2016. Έχουμε τη διτή τάση να χρηματοδοτούμε και μικρά και μεγάλα έργα. Θέλουμε να χρηματοδοτούμε μικρά project, Όμως διοικητικά είναι πιο εύκολη η χρηματοδότηση πιο μεγάλων έργων. Όμως, όταν βλέπουμε τι πραγματικά υλοποιείται και τι πραγματικά απευθύνεται στον πολίτη και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, αυτό το έργο είναι πάντοτε μικρό. Και είναι σημαντικό να χρηματοδοτούμε και αυτά τα μικρά έργα και ε, λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό το κριτήριο όταν αποφασίζουμε δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, να σας υπενθυμίσω ότι από το... 2016 ξεκινά να λειτουργεί και το νέο Ταμείο Εγγυήσεων, το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει εξηγήσει. Ή μάλλον διορθώνω. Η δική μας Επιτροπή θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξηγήσει για το μοντέλο που θα ακολουθηθεί. Θέλετε να παρέμβετε. Όχι. Άρα να κάνουμε μια διακοπή 5 λεπτών, περιμένοντας να έρθει Περιμένοντας να έρθει ο Επίτροπος βράψεις. Πέντε λεπτά διακόπη παρακαλώ. Ναι, διακοπή 6-7 λεπτών. Μέχρι να έρθουν οι συνάδελφοι αρμόδιοι ε, και ο φιλανδός συνάδελφος ο εισηγητής ε, από πλευράς Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού. Διακοπή 5 6 λεπτών, τα λέμε εντός ολίγου. No, il collega Fernandez che è un po' in ritardo, scusateci. Όχι, ζητώ συγγνώμη, ο συνάδελφος Φερνάντες είναι που έχει καθυστερήσει, που είναι δικό μας, δικός μας συνάδελφος. Η διακοπή παραμένει όμως.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 Συνάδελφοι, φτάνει ο κύριος Φερνάντες, όπου να είναι. Merci Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Κύριε Φερνάντες. Ακούσαμε προηγουμένως τον συνάδελφο Σδρογεύσκη που είναι εδώ και, ήταν, και είναι εισηγητής μας για τον προπολογισμό του 2016. έκθεση του έχει σχέση και με το δικό, δικό σας έργο. Ακούσαμε προηγουμένως ποιες είναι οι προτεραιότητες των συναδέλφων για το 2016 και ξέρουμε ότι εσείς βαδίζετε σε αυτόν τον ε, δρόμο, την πορεία συναντήσεων με τις επιτροπές. Πρέπει να είμαστε η δέκατη επιτροπή που συναντάτε και ξέρετε ότι οι γενικές και στατικές προτεραιότητες της Επιτροπής μας και των υπόλοιπων επιτροπών είναι κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. η κεντρική σημασία της εκπαίδευσης ε, και του πολιτισμού ε, στις δεξιότητες, της τεχνολογίας, στις πολιτικές για τους νέους, στην πολιτική για τους πολίτες και το οπτικοακουστικό σύστημα και ο αθλητισμός είναι αρμοδιότητες μας και είναι θέματα που έχουν όλο ένα μεγαλύτερη σημασία στην Ευρώπη που αναπτύσσεται και θέλει να ε, εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων όντας βιώσιμη και ευφύς. Σε αυτή τη φάση να σας δώσω αμέσως το λόγο και μετά στον συνάδελφο Σντρογεύσκη, αλλά και σε όσους συναδέλφους θέλουν να συμμετάσχουν. Είναι σημαντικό να έχουμε μια σφαιρική εικόνα για τον προπολογισμό και να δούμε το θέμα των πληρωμών, καθότι το Κοινοβούλιο έχει δώσει αγώνα για το θέμα αυτό. Το θέμα των προτεραιοτήτων, και το να δούμε πώς ο προπολογισμός του 2016 μπορεί να συνδυαστεί με το επενδυτικό πρόγραμμα Juncker. Να ε, ενεργοποιήσουμε δηλαδή μια εταιρική σχέση που να είναι εξαιρετικά σημαντική. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη. Καθυστέρησα γιατί υπήρξε μια άλλη καθυστέρηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και είχα εγγραφεί για να θέσω ερώτηση προς τον κύριο Ντράγκη. Χρειάστηκε λοιπόν να περιμένω οιμέ και γι' αυτό καθυστέρησα και θα πρέπει να ε, ζητήσω συγγνώμη. Ε, να σας ευχαριστήσω, έρχομαι εδώ περισσότερο για να ενημερώσω, αλλά πάνω απ' όλα για να καταγράψω τις δικές σας μέρημνες. Ήδη έχουμε γκρίνει κατευθυντήρια γραμμή για τον προϋπολογισμό την Ολομέλεια του Μαρτίου, προτεραιότητα για την απασχόληση, το πνεύμα του επιχειρήν, τις ε, προτεραιότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα 3 ε, την εσωτερική αλληλεγγύη, την εξωτερική αλληλεγγύη, την ασφάλεια, την μετανάστευση και άλλες προτεραιότητες. Ξεκινούμε από την αρχή ότι σεβόμαστε τις δεσμεύσεις μας και τις συμφωνίες που έχουν ε, συναυθεί. Ως προς τις πληρωμές υπήρχε συμφωνία για να μειωθεί το ποσό των ε, μη κατευθύντων ποσών από το 2013 2016 σε ένα μέγιστο ποσό 2 δις για το 2016. Όμως ε, αυτό το πρόβλημα ελπίζουμε να βρει οροστική λύση και κάποια στιγμή να πληρώσουμε αυτά που πρέπει, γιατί οι πληρωμές είναι αναγκαστική συνέπεια των ε, δεσμεύσεων των αλήψεων πιστώσεων. Ε, για το πρόγραμμα Juncker τώρα, για το Ευρωπαϊκό Στατικικό Ταμείο, για τα περιθώρια που δεν θα χρησιμοποιηθούν, να πω ότι μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε από το 2016. Αυτή είναι η ευελιξία που θελήσαμε. Η ευελιξία λοιπόν αυτή είναι σημαντική. Το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 το αποδεχτήκαμε γιατί ακριβώ είχαμε τη δυνατότητα αξιοποίηση αυτών των περιθωρίων. Και κατά την αξιοποίησή του θα πρέπει αυτό να το θυμίζουμε διαρκώ καθώ και τα υπόλοιπα εργαλεία ευελιξία που διαθέτουμε. Για το χρονοδιάγραμμα να σα πω ότι θα εγκρίνουμε στις 23 Ιουνίου στην Επιτροπή την εντολή για τους τριμερείς διαλόγους και στην Ολομέλεια τον Ιούλιο και πάλι την εντολή στις 3 Σεπτεμβρίου προθεσμία υποβολή τροπολογιών για τον προπολογισμό από τις Επιτροπές ή από τους βουλευτές, 10 Σεπτεμβρίου για τις πολιτικές ομάδες, ε, μέσα Σεπτεμβρίου έγκριση από τον Πενευτικό Προπολογισμό για την έκθεση με ψήφισμα τον Οκτώβριο, 29-30 Σεπτεμβρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών για τις ε, τροπολογίες, 12-13 Οκτωβρίου ψηφίζουμε για, το, για την έκθεση, τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια και τον Νοέμβριο στην Διαλλαγή. 27 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιο έκθεσης μπορώ να πω ότι συνολικά είμαστε ικανοποιημένοι, ελπίζω και η Επιτροπή ε, Πολιτισμού, συγγνώμη, το Erasmus ΣΥΝ, σε αυτό το σχέδιο προπολογισμού, έχει αύξηση ως τις αναλήψεις 7,4% σε σχέση με το 2015 και για τις πληρωμές 30,1%. Και πάλι σε σχέση με το 2015. 75% των πληρωμών αφορούν τι αναλήψει του 2016 και μόνο 25% είναι για να πληρωθούν τα μη καταβληθέντα. Για να το πω έτσι. Για το κεφάλαιο 3. Δεν υπάρχει περιθώριο Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το εργαλείο ε, ευελιξίας, 124 εκατομμύρια νομίζω είναι. Θα δούμε λοιπόν εδώ ε, τι θα αξιοποιήσουμε. Τα προγράμματα της Κούλτ, όπως η Ευρώπη της Δημιουργίας, έχουν αύξηση των αναλήψεων 8%, σε πληρωμές 18,7%, η Ευρώπη για τους πολίτες αύξηση 4,5% και για τις πληρωμές 29,9%. Για τις δράσεις επικοινωνίας επίσης αύξηση και αυτές ήταν οι σημαντικότερες πληροφορίες. Υπάρχουν επίση τα πιλωτικά προγράμματα και παρασκευαστικέ δράσει. Εκεί δεν έχουμε περιθώριο, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αξιοποιήσουμε τι δυνατότητε ευελιξία για το στόχο αυτό. Θεωρούμε ότι τα πολυπιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικέ δράσει είναι σημαντικά. Και στόχος μας είναι να τα προασπίσουμε. Και κάτι ακόμα. Όταν έγινε το front loading της πρωτοβουλίας για τους νέους 2014-2015, το 2016 δεν είχαμε δεσμεύσεις. Και θέλουμε αυτό το πρόγραμμα να συνεχιστεί. Πολλοί συνάδελφοι δεν είδαν ακόμα και δεν το πρόσεξαν ότι το 2016 δεν υπάρχουν commitments, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για την ε, πρωτοβουλία για τους νέους. Γιατί είχε γίνει το front loading, τα 6 δις ευρώ 2014-2015. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε ήδη από την εντολή για τον τριμερείς διαλόγους και θα είναι προτεραιότητα που δεν θα είναι εύκολη, μια από τις πρώτες προτεραιότητες για την απασχόληση είναι να έχουμε ευελιξία. Να εγγράψουμε τα ε, αχρησιμοποιητά περιθώρια για το στόχο αυτό και να έχουμε δεσμεύσεις, αναλήψεις για το 2016. Θέλουμε τέτοιες δεσμεύσεις για το 2016 για το πρόγραμμα αυτό που είναι σημαντικό. Βεβαίως εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Το ποσοστό ενέργεια είναι υψηλότατο, ιδίως για τους νέους. Αλλά υπάρχουν και πολλά κονδύλια που δεν χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με αυτό, πώς πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες. Πάντως, είναι κάτι που συνεχίζει να είναι προτεραιότητα. Το πιστεύω, αλλά θέλω να σας ακούσω κιόλας, να ακούσω τις απόψεις σας. Αυτές τις γρήγορες πληροφορίες ήθελα να σας δώσω, αλλά όπως έλεγα, κυρίως θέλω να γνωρίζω ποιες είναι οι δικές σας μέρημνες, οι δικές σας προτεραιότητες και οι δικές σας επικρίσεις ενδεχομένως, για να μπορέσουμε να έχουμε τον καλύτερο δυνατό προϋπολογισμό. Γι' αυτό ήρθα. Σας ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη ενημέρωση, ο λόγο του συνάδελφου Στρογεύσκη, διότι είναι υπεύθυνο για τον προπολογισμό. Μετά και στου συναδέλφου θα τη ζητήσουν. Αλλά να πούμε ότι σε αυτή την επιτροπή συζητήσαμε μακρόν όπω και σε όλο το κοινοβούλιο, το τι θέλουμε για το 2014-2020 με σοβαρά περιθώρια για το Erasmus ΣΥΝ, την Ευρώπη τη Δημιουργία. Και οι αιτήσει αυτέ αυξήσει έχουν να κάνουν με όσα προγραμματίζονταν ούτω ή άλλω. Ενώ για την Ευρώπη των πολιτών το συζητήσαμε και προηγουμένω με τον Επιτροπό Αβραμόπουλο, Όντω υπάρχει μια μικρή αύξηση, αλλά έτσι κι αλλιώ υπήρχε ραχική μείωση του 14%. Πάλι είμαστε κάτω από το όριο το αρχικό και αυτό επίσης που μας απασχολούσε πολύ είναι η πρωτοβουλία για τους νέους, γιατί υπάρχει και η διάσταση της εκπαίδευσης, ε, την αγγίζει η πρωτοβουλία των νέων και γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς να πω το εξής. Γενικά όλη η χρηματοδότηση του πολιτισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Το πιο εύκολο λοιπόν θα ήταν να πούμε εντάξει ας αφήσουμε την Επιτροπή Πολιτισμού να έχει αυτά που έχει γιατί ούτως ή άλλως δεν σημαίνει και πολλά μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο. Το λέω αυτό γιατί κάθε χρόνο γίνονται παρεμβάσεις ας πούμε στην γεωργική αγορά ε, που είναι ε, πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είναι ε, σε συνδυασμό οι δαπάνες για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά χρειάζεται να βρούμε περισσότερα χρήματα για τον πολιτισμό, καθώς είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Για να μπω τώρα σε λεπτομέρειες. Καταρχάς χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το Erasmus Plus έλαβε μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Συνεχώς λέμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, είναι μεγάλη η αξία του. Πραγματικά θέλουμε μια ισορροπημένη κατάσταση έτσι ώστε οι δεσμεύσεις του παρελθόντος να μην ε, φάνε όλα τα χρήματα που ε, ε, έχουμε λάβει επιπλέον. Ό,τι τέλος πάντων υπάρχει σε επίπεδο χρηματοδότησης πρέπει να προστατευτεί. Ενδιαφερόμαστε επίσης πάρα πολύ για το Euronet Plus. Τι συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Αυτό το πρόγραμμα θα έπρεπε να έχει εγγύηση σε τριετής. Όμως η διαδικασία σταμάτησε και τώρα μας έχουν υποσχεθεί 5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά τουλάχιστον το 1 εκατομμύριο ε, είναι, είναι τουλάχιστον 1 εκατομμύριο λιγότερο από ό,τι μας είχαν υποσχεθεί αρχικά. Και υπάρχει και το πρόβλημα με τις προθεσμίες. Ε, βέβαια, αν εμεί έχουμε προβλήματα με προθεσμίες, τότε εσείς κύριε Φερνάντες έχετε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί πολλές φορές η διαδικασία είναι πολύ σύντομη, άλλε τρέχει παράλληλα. Πρακτικά λοιπόν ο χρόνος δράσης είναι περιορισμένος. Αυτό αφορά στα πιλωτικά έργα. Εμείς πρώτα θα ψηφίσουμε και μετά ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα λάβουν υπόψη αυτά που ψηφίσουμε. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Είναι λίγο αντίστροφη πλέον η διαδικασία. Τώρα για τη χρηματοδότηση των προπαρασκευαστικών δράσεων και των πολιτικών έργων. Αυτό θα είναι το περιθώριο που έχουμε τώρα, θα διορθωθεί στο μέλλον. Τι κονδύλια θα δώσει η Κομισιόν. γιατί υπάρχουν ε, πολλές δυσκολίες στο οικονομικό πεδίο. Έλαβα πληροφορίες από την γραμματεία που λένε ότι τα πιλωτικά έργα δεν θα λάβουν πλέον χρήματα. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν όντω ισχύει αυτό. Τώρα οι υπόλοιποι συνάδελφοι, η συνάδελφος ε, Φερνάιεν. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς ε, που ε, αφιερώσατε χρόνο για να έρθετε εδώ και να συζητήσετε μαζί μας σημαντικά ζητήματα για τον πολιτισμό. Είχαμε και μία εντατική συζήτηση με τον Επίτροπο Αβραμόπουλο για το πρόγραμμα για τους πολίτες. Ε, τη τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η τάση να τελειώνει ο προϋπολογισμός στα μεγάλα εμβληματικά έργα και να μένει πολύ μικρό κομμάτι του προϋπολογισμού που είναι πιο μικρά. Δηλαδή αυτά που είναι 5, 6, 7 εταίροι έχουν μεγαλύτερη τύχη από ότι τα μικρότερα project που τελικά προσφέρουν περισσότερα στην Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και σχετίζεται με τον προϋπολογισμό. Πρέπει να γράφεται και στον προϋπολογισμό. Για το Euronet Sin, εδώ και πολλά χρόνια υπήρξε μία μόνιμη χρηματοδότηση. Κάθε χρόνο υπήρχαν νέες αιτήσει για αυτό το δίκτυο των ραδιοφωνικών σταθμών και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είμαστε ένα κοινό μέτωπο και να λέμε ότι πραγματικά είναι αντιπαραγωγικό να μην υπάρχει μία συνεχής χρηματοδότηση αυτού του δικτύου δεν είναι να δώσεις λεφτά για ένα χρόνο, πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Νομίζω ότι είναι σημαντικό επίσης να γίνει ξεκάθαρο ότι στα πλαίσια του προγράμματος επενδύσεων που κατέθεσε ο Γιούνκερ πρέπει να υπάρχουν και μέτρα ε, για τον πολιτισμό συγκεκριμένα για την βιομηχανία του πολιτισμού και την εκπαίδευση. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο αυτά πρέπει κατά τη γνώμη μου οι επενδύσεις να ανήκουν και αυτές στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης γιατί η οικονομική ανάπτυξη, το οικονομικό δυναμικό ε, καλλιεργούνται μέσα από αυτό ε, και οι επενδύσεις στην ε, εκπαίδευση στην ουσία πρέπει να υποστηρίζονται συνεχώς έτσι ώστε να έχουμε προσωπικό με σωστά προσόντα για να είναι και ανταγωνιστικό. Αυτό ε, μπορεί να γίνει με την υποστήριξη των ετοιμάτων που έχουμε εμείς καταθέσει εδώ από το Κοινοβούλιο με τις τροπολογίες μας γιατί πραγματικά πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μα ότι η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική για την ε, περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ η Γερτρούδη. Ευχαριστώ κύριε Φερνάντες που είστε μαζί μας και για τη συνεισφορά σα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο πολιτισμός, ε, η πολιτισμική οι ανταλλαγές σε επίπεδο πολιτισμού και ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι η ακρογωνία, είναι η της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν μπορεί ο κόσμος να έρθει σε επαφή, ε, δεν είναι εύκολο ένας να σέβεται τον άλλον. Είναι σημαντικό λοιπόν στοιχείο της Επιτροπής αυτής αυτό το θέμα και είναι σημαντικό και για την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Υποστηρίζω αυτά που ήδη υπόθηκαν ότι ε, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα πρέπει η εκπαίδευση και ο πολιτισμός να αποτελούν σημείο ε, στο οποίο θα δοθεί μεγάλη ε, έμφαση για να έχουμε την κατάλληλη εξέλιξη τα επόμενα χρόνια. Για το ΣΥΝ έχουμε αύξηση του προϋπολογισμού κατά 40% μέσα στα πλαίσια του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Όμως αυτό είναι κάτι που το είχαμε ε, που το περιμέναμε, αλλά δεν αρκεί για τις ανάγκες των κοινωνιών μας. Αν υπάρχουν λοιπόν οποιασδήποτε δυνατότητες για αλλαγή του βάζου προπολογισμού προς τη δική μας ε, αρμοδιότητα θα θέλαμε να ε, γίνει. Μιλήσατε επίσης προηγουμένως για τις αυξήσεις ε, που όμως δεν αρκούν και ήταν ξεκάθαρο όταν μιλήσαμε προηγουμένως με τον ε, Επίτροπο ότι πολλά έργα απορρίπτονται. Δεν υπάρχει διαφήμιση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. υπάρχουν πολλοί κόσμοι που θα ήθελε να εμπλακεί και δεν το κάνει. Άρα πρέπει να γίνουν περισσότερα τα επόμενα χρόνια για να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερο προϋπολογισμό στο ε, πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες, κάτι παραπάνω από αυτό που έχει. Και κατ' εμέ το πρόγραμμα Euronet Plus Χρειάζεται και αυτό επιπλέον κονδύλια και πρέπει να συνεργαστούμε γι' αυτό γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή η επικοινωνία μέσα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα δίκτυα που φτάνουν στον κάθε ένα πολίτη είναι ο πιο καλός τρόπος για να μιλήσουμε για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Μόργανο. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε για την ε, παρουσία σας. Είναι σημαντικό για να ακουστούν κάποιες προτηρήσει. Θέλω να υπογραμμίσω δύο πτυχές και σε συμφωνία μας είπαν οι συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα η σχέση μεταξύ της αύξησης των ε, δεσμεύσεων για τις διάφορες επιμέρους γραμμές χρηματοδότησης που αφορούν την, τον πολιτισμό και την αύξηση των πληρωμών και τους αριθμούς που γνωρίζετε. Και το δεύτερο, ε, αυτό που είναι πολύ σημαντικό νομίζω είναι οι προκαταβολές ε, και σε σχέση με το πώς προηγουμένως έχει εκτελεστεί ο προπολογισμό, αλλά και το πώς μπορούμε να διαθέτουμε ε, τα ποσά. Διότι αυτό έχει σχέση με το κατά πόσον θα υπάρχει βεβαιότητα. Γι' αυτό κάνω αυτή την αναφορά και γιατί αληθεύει ότι αν τα μέτρα για ένα πλαίσιο παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται ανάλογα με τις δεσμεύσεις τα κονδύλια του πολιτισμού φαίνεται να είναι κάτι που περιθωριακά απασχολεί ως προτεραιότητα. Και έρχεται ο πολιτισμός να καλύψει το χάσμα μεταξύ της αντίληψης των πολιτών σε σχέση με την ε, ίδια την Ένωση και το τι θα πρέπει να υλοποιηθεί. Έτσι λοιπόν δεν είναι συνδικαλιστική η δική μα επιδίωξη το να δοθεί έμφαση στον πολιτισμό, απλώ πρέπει να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο και από αυτή την διαρκή αμφισημία. Και το λέω και σε σχέση με την άλλη πολύ σημαντική διάσταση που και εσεί εντοπίσατε. Δηλαδή, ευτυχώ δόθηκε προτεραιότητα στην απασχόληση και αυτό θα μα έλειπε. Όμω, και ο πολιτισμό είναι σε θέση να δώσει μια σοβαρή απόκριση στα θέματα τη απασχόληση. Συνολικά λοιπόν και για να μην μακρηγορώ. Αναφερθήκατε και στα πιλωτικά προγράμματα. Νομίζω ότι είπατε πόσο σημαντικά είναι και θα συμφωνήσουμε. Όμως με την κατάσταση ως έχει, ε, αναρωτιέται κανείς τι θα γίνει με τη διάθεση των ποσών και με τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Θέλαμε ως προς αυτά να καταλάβουμε κάποια περισσότερα. Γιατί νομίζω τα δύο θέματα είναι λένε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Να προσθέσω το εξής όσα υπόθηκαν. Ότι ποιος λέει Α, δεν σας έδραζα το λόγο, παρακαλώ. Η κυρία Κάμερφερτ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ συντάσσομαι και υπογραμμίζω όλα όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Ε, απλώς υπάρχουν δύο στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά. Ε, υπάρχουν πολύ περισσότεροι που καταλαβαίνουν το προπολογισμό καλύτερα από μένα, όμως αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι αυτό που είπε και ο συνάδελφος στο Γεύση. Έχουμε τρία προγράμματα για τα οποία έχουμε τόσο λίγα χρήματα που στην ουσία δεν επιτρέπεται ε, σε οποιαδήποτε θέση να να κάνουμε αυτό το οποίο μας έχουν υποσχεθεί μέσα στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού ε, προγράμματος. Είναι τόσο σημαντικά αυτά τα προγράμματα και υπάρχει συνένεση τελικά ότι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δεχτούμε να υπάρχουν τόσο λίγα κονδύλια. Επίσης είναι επίγον ε, αυτό το θέμα μεταξύ πιστώσεων, πληρωμών και πιστώσεων ε, υποχρεώσεων, ειδικά για το Erasmus Plan, ε, Plus, να ε, λυθεί. διότι για το Erasmus ειδικότερα, για τις υποτροφίες, δηλαδή για τους φοιτητές, φέτος τον Ιούλιο δεν θα έχουμε πια χρήματα. Και το 2016 δεν θα αλλάξει η κατάσταση. Αυτά είναι πράγματα ορατά ε, που δείχνουν προς τα έξω την Ευρώπη αυτά που κάνουμε μέσα από το Erasmus Plus ε, πάνε στους πολίτες κατευθείαν και αν δεν γίνουν οι πληρωμές ε, μας λείπει σημαντικό κομμάτι της ορατότητας της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό πρέπει επιγόντως να προσέξουμε το Erasmus Plus να γίνουν οι πληρωμές. Επίσης για το Euronet Plus να υπογραμμίσω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι γιατί και από την πλευρά μου κατέθεσα τροπολογία και θεωρώ ότι πρέπει επιγόντας να συζητήσουμε τι θα κάνουμε στο μέλλον με το Euronews. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα πρόβλημα περιεχομένου και αν υπάρχουν χρήματα από κάπου να τα πάρουμε και να γίνει εξοικονόμηση από κάπου αλλού, είναι πολύ σημαντικό να δοθούν στο Euronews γιατί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ειδικότερα όσον αφορά στην ιδιωτική χρηματοδότηση η οποία γίνεται όλο και περισσότερο μέσα από το μέσω του Euronews και πραγματικά δεν ξέρω, πρέπει να το συζητήσουμε αν ε, πρέπει να ε, το υποστηρίξουμε κάπως αλλιώς γιατί δεν θα έχουμε τελικά ανεξάρτητη δημοσιογραφία έτσι. Πέτρα και Λουέρτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι συμφωνώ απολύτως με την Πέτρα ως προς το Euronet και το Euronews. Η θέση μας στο ECR είναι κάπως διαφορετική από αυτή των άλλων συναδέλφων. Εμείς δεν θέλουμε μόνο απλά περισσότερα χρήματα και πιστεύουμε ότι τα 25 εκατομμύρια ευρώ που παίρνει το Euronews ως επιδότηση είναι κάτι που δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάστηκε 8 εβδομάδες για να απαντήσει στο κοινοβουλευτικό ερώτημα που κατέθεσα. Ε, τεράστια καθυστέρηση εκτός ε, προβλεπόμενου χρόνου και καταδέχθηκε να μου απαντήσει κατά σύμπτωση την ίδια μέρα κατά την οποία δημοσίευσα στον τύπο το παράπονό μου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μου απαντάει. Πρέπει να σεβαστούμε τα ισχύοντα. Εγώ δεν είμαι υπέρ των επιδοτήσεων στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά εν πάση περιπτώσει αν πρόκειται να έχουμε τέτοιου είδους στήριξη, να τις έχουμε για ανεξάρτητους φορείς επικοινωνίας και όχι για το Euronews. Δεν πιστεύουμε ως συντηρητικοί μεταρρυθμιστές ότι πάντοτε είναι καλύτερη η περισσότερη δαπάνη, η αύξηση των δαπανών και η μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τεκτενόμενα της ζωής του Ευρωπαίου πολίτη. Θεωρούμε όμως ότι μπορεί η Ευρώπη να συμβάλλει και να έχει προστιθέμενη αξία π.χ. στο Erasmus Plus, στο ΣΥΝ ή στην έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Τέτοιου είδου μηνύματα όπω αυτά που ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βοηθούν καθόλου τους Βρετανούς πολίτε ε, οι οποίοι θέλουν όλο και περισσότερο να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρομαι στο θέμα τη Ευρωπαϊκή Εθαγένεια μεταξύ άλλων. Ίσως δεν είναι η πιο σωστή προσέγγιση. Εμεί θέλουμε, εγώ προσωπικά θέλω να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να τεθεί συζήτηση σε μια κάπως διαφορετική βάση και να μην έχουμε μόνο υψηλότερε δημόσιες δαπάνες και να μην θεωρείτε ότι αυτό είναι εγγενώς καλό, να θεωρηθεί ότι οι ψηλότερες δημόσιες δαπάνες είτε από Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από κράτη-μέλη είναι καλές όταν είναι στοχευμένες εκεί που πραγματικά υπάρχει ένα ανάγκη. Ευχαριστώ. Να θυμίσω ότι η χώρα σας είναι από αυτές που λίγο που περισσότερο ωφελούνται από το Erasmus είναι. Έχει μεγάλο ποσοστό από τη χρηματοδότηση γιατί έτσι το έχει ζητήσει. Και κυρία το ζήτησε. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήτης, να πω ότι εμείς δεν θέλουμε περισσότερα χρήματα για το Euronews. Θέλουμε ε, όμως ε, μια ε, συνεχή ε, υποστήριξη του Euronet. Δεν ξέρω αν μέσα από την μετάφραση πραγματικά τα καταλάβετε διαφορετικά, αλλά το Euronet Plus είναι στην ουσία ε, μια, ε, ένα συνεταιρισμός μικρών τοπικών ε, ραδιοφωνικών σταθμών που χρειάζονται υποστήριξη γιατί τελείως δεν μπορούν να, να κάνουν παραγωγές. Αυτό είναι μόνο ε, προς το συμφέρον ε, έχει προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη να δίνονται δηλαδή χρήματα και κονδύλια ε, σε μικρούς σταθμούς που δεν έχουν ίδια μέσα και αυτό πραγματικά συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει για τις μικρές επιχειρήσεις. Όμως για το Euronews Εκεί που υπάρχουν εκατομμύρια επενδύσεις και μεγάλοι επενδυτές, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται να μπαίνει με τόσα χρήματα. Πραγματικά και εγώ θα ήμουν υπέρ του να κοπούν χρήματα από το Euronews και να πάνε στο Euronet Plus. Ε, πολύ εύκολα. Πραγματικά καλό θα είναι να δούμε, να ελέγξουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο θέμα του Euronews σε επίπεδο ε, Ουκρανίας, σε επίπεδο ε, ιδιωτών επενδυτών, να δούμε τι συμβαίνει. Από άποψη λοιπόν Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Euronet Plus όμως, για αυτό το συνεταιρισμό των ραδιοφωνικών σταθμών, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει η χρηματοδότηση. Ευχαριστούμε για αυτές τις διευκρινήσεις και συμφωνώ για αυτή, με αυτή τη διάκριση. Το Euronet είναι ένα δίκτυο που χάρη σε αυτά τα κονδύλια που είναι σημαντικά καταφέρνει να δίνει σοβαρότητες ειδήσει για την ε, Ευρώπη και ανεξάρτητα διόφωνα και το καθεξής. Το Euronews είναι κάτι διαφορετικό, είναι όμως θέμα πολύ ευαίσθητο και ίσως καλύτερα να εμβαθύνει η Επιτροπή Πολιτισμού. Θα το συζητήσω εντός λίγο με τους συντονιστές. Θα προβλέψουμε περαιτέρω συζήτηση για τα θέματα αυτά, είτε μιλάμε για το Euronews, Europeana και Euronet. Είναι όλα σχετικά με την επικοινωνία που θα μας απασχολήσει και πρέπει να εμβαθύνουμε γιατί όντως προβλήματα υπάρχουν. Αυτά είναι ελλείμματα του προπολογισμού. Με κάποιε ιδιαιτερότητε να προσθέσω κάτι μόνο. Ο πολιτισμός δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Μιλάμε για παιδεία, μιλάμε για ενημέρωση, μιλάμε για το ΑΕΠ της Ευρώπης και ίσως να μην είναι γνωστό αυτό. Οι βιομηχανίες της επικοινωνίας η, η πνευματική δημιουργία είναι σημαντικό κεφάλαιο για την Ευρώπη. Είναι 50% τη ευρωπαϊκή οικονομία. Υπάρχει λοιπόν και πολιτισμό στον προπολογισμό και η ευρωπαϊκή πολιτιστική κοινωνία πρέπει να προστατευτεί και η ψηφιοποίηση πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο πολιτισμό έχει σημασία στον διαπολιτισμικό διάλογο και όλα αυτά οδηγούν την Ευρώπη στην ανάπτυξη. Υπ' αυτήν την έννοια πρέπει να επιμείνουμε τα θέματα αυτά, πρέπει να ε, διατηρήσουν την κεντρική του σημασία και σε τη διαστολή με την εγγύηση για τους νέους, ε, τα προγράμματα αυτά και το Erasmus Sin και η Ευρώπη της Δημιουργίας δεν ε, οδηγούν σε κατασπαρτάληση κανενός ευρώ, ούτε ενός. Όλα τα κονδύλια αξιοποιούνται, εξαντλούνται και αξιοποιούνται. Επίσης, εφόσον υπάρχει ζήτηση μεγαλύτερη ε, από ό,τι προβλέπουμε, καλό είναι να σκεφτούμε ότι ο στόχος είναι να ικανοποιούνται οι ανάγκες των ε, όσων μας ζητούν να λάβουμε δράση. Σας ευχαριστώ και σας δίνω το λόγο για να κλείσετε. Ευχαριστώ όλους και όλες. Σας διαβεβαιώ ότι μπροστά σας έχετε ένα σύμμαχο. Είμαι σύμμαχό σας, φιλόδοξος και ρεαλιστής συνάμα. Την ίδια φιλοδοξία είχαμε όταν ασχοληθήκαμε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Όλοι έλεγαν ότι είναι αδύνατο να μειωθούν οι περικοπές για, στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2006 και στο πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη. Και όμως τα καταφέραμε κατά ένα δις. Και αυτό για τον προπολογισμό το 2016 θα έχει θετικές επιπτώσεις και θα προσπαθήσουμε να του ξαναδώσουμε το προπολογισμό του 2016 το, τα χρήματα που του είχαμε πάρει. Μιλάμε για 145 δις ευρώ για ε, το 2016, αλλά το 6% αυτών έχει να κάνει με τις διοικητικές δαπάνες και δαπάνες λειτουργίας. Άρα 84% θα πάει στις επενδύσεις. Καμία χώρα δεν ξέρω όπου οι διοικητικές και οι λειτουργικές δαπάνες να είναι μόνο το 6% του προϋπολογισμού. Αυτό το νούμερο αναδεικνύει τη σημασία του προϋπολογισμού Αποδεικνύει επίσης την προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού και στην πολιτική για την νεότητα, για τους νέους για παράδειγμα ή για τον πολιτισμό ή και για την εκπαίδευση αν θέλετε. Αυτά είναι ε, στο πεδίο της εθνικής αρμοδιότητας κάθε κράτους μέλους. Ωστόσο ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει σε πολλά κράτη-μέλη περισσότερα από ότι ο εθνικός τους προϋπολογισμός για την άσκηση τέτοιου είδους πολιτικής. Υπάρχουν κάποια όρια δημοσιονομικά, κάποια όρια στον προϋπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει αυτή την πρόταση. Θα δούμε ποια ανάγνωση θα της επιφυλάξει το Συμβούλιο. Και θα δούμε επίσης τι πρέπει να γίνει για να έχουμε τη φιλοδοξία που τόσο μου αρέσει αλλά και τον ρεαλισμό που είναι απαραίτητος στα πιλωτικά προγράμματα, στις προπαρασκευαστικές δράσεις γιατί στον οικονομικό κανονισμό ε, προβλέπεται ότι μόνο 140 εκατομμύρια θα έχουμε, λέει ο μιλητής. Όμως το τρίτο τίτλο δεν έχουμε καθόλου περιθώριο για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Τι είναι σαφές για την εντολή που έχουμε για τον τριμερή διάλογο. Ε, λοιπόν, θέλουμε να αξιοποιήσουμε την ευελιξία, την ευελιξία για να αυξήσουμε τα περιθώρια, για να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη δράση, μεγαλύτερο πεδίο δράσης για τις προπαρασκευαστικές δράσεις και για τα πιλωτικά προγράμματα στον τίτλο 3. Έχουμε τέτοιο περιθώριο στον τίτλο 1, αλλά δεν το έχουμε στον τίτλο 3 και πρέπει να έχουμε την ευελιξία για να το πετύχουμε αυτό το περιθώριο και μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα χρηματοδοτικά μέσα ευελιξίας. Το Erasmus Συν, το Erasmus Plus το αυξήσαμε κατά 40%, 40,5% 14,7 ε, δις ευρώ που πήραμε από το 2011, το αυξήσαμε για τα έτη 14 με 17 και αυξήσαμε και τις δεσμεύσεις 15 με 16 εκατομμύρια για το 2015 και αυτό θα έχει επίπτωση στις πληρωμές. Πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι ε, αρκετά χρήματα για τις πληρωμές. Αυτά λοιπόν για τα πιλωτικά project και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Βασίζομαι στη βοήθειά σας για να υπάρξει ευελιξία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Με πείθει ιδιαίτερο στο επιχείρημα ότι ο τίτλος 3 στον προϋπολογισμό έχει μικρότερο ειδικό βάρος από τους άλλους δύο τίτλους ή τους υπολείπους εν πάση περιπτώσει. Το δέχομαι αυτό, επομένως μια αύξηση κατά μεγάλο ποσοστό ενός μικρού τίτλου είναι μικρότερη από μια μικρότερη ποσοστιαία αύξηση αλλά κονδυλίων που βρίσκονται σε ένα τίτλο άλλων και όχι των τρία όπου τα μεγέθη είναι ε, αυξημένη. Βεβαίως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση είναι εξαιρετικά σημαντικά θέματα αλλά εξίσου σημαντικό είναι και η ενημέρωση, η πληροφορία. Πρέπει να αξιοποιούμε σωστά τα προγράμματα που βρίσκονται στη διάθεσή μας. Γνωρίζω πολύ καλά τα προγράμματα για τους νέους, για τον πολιτισμό, για την εκπαίδευση, γιατί στη χώρα μου έχω γράψει ένα βιβλίο που περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα για την εκπαίδευση, για τα νιάτα, για τον πολιτισμό, που, όλα τα προγράμματα που είναι διαθέσιμα και ε, αυτό δείχνει την Ευρώπη χωρίς σύνορα. Τώρα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. είναι ανοιχτό για επενδύσεις για τον πολιτισμό και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Μιλήσαμε για τις προτεραιότητες. Και είναι σημαντικό για να ξέρουμε εάν τελικά πρέπει να κάνουμε redeployment, δηλαδή να πάρουμε τα χρήματα από μία γραμμή του προϋπολογισμού και να τα βάλουμε σε άλλη. Και σημειώνω και το ερώτημα για το Euronet Plus, το SIN, το Euronet SIN, το σημειώνω και στη συνέχεια θα δούμε ξανά αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού. Ελπίζω το Συμβούλιο να αναγνώσει με καλό τρόπο τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό, γιατί ξέρετε, ε, συχνά από εγώ βόμαστε. Λέμε ότι πρέπει να σεβαστούν τις δεσμεύσεις, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρέπει να σεβαστεί το Συμβούλιο τις, ε, τους συμβιβασμούς και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Αλλά πρέπει και κυρίως να σεβαστεί τις ίδιες τις δημόσιες δηλώσεις που έχει κάνει το Συμβούλιο. Και όλα αυτά συμβάλλουν στην απασχόληση που είναι η προτεραιότητα την οποία υπερασπιζόμαστε εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Υπολογίζουμε στη στήριξή σας εφόσον εκδώσατε, έχετε δημοσιεύσει και αυτό το βιβλίο. Να θυμίσω στους συναδέλφους ότι 30 Ιουνίου είναι η προθεσμία. Σας χαιρετούμε και περνάμε απευθείας στις συνεδρίες των συντονιστών γιατί έχουμε αργήσει κάπως.